Everybody to... Παρακαλώ όλες και όλους καθίστε. Can I welcome you to the meeting this morning? I have uh, just a few Σας καλωσορίζω. Πρώτα λίγες ανακοινώσεις. Η ε, σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται ηλεκτρονικά. Είναι στο λεγόμενο web stream, να το έχετε υπόψη σε αυτό. Δεύτερο, λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις εχθές στη συνάντηση των συντονιστών, τις οποίες θα σας διανύμουμε. Και αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν έχετε προβάλει ενστάσεις, τότε θα θεωρηθούν εγκεκριμένες. Και επίσης ρωτώ αν όλες και όλοι έχετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας, διότι ίσως σήμερα να γίνουν κάποιες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Ας προχωρήσουμε τώρα στο υπαριθμόν 7, προϋπολογισμός 2010, τμήμα 3, Επιτροπή. Ε, και μιλούμε για τη γνωμοδότηση για την διαδικασία του προϋπολογισμού και για το τμήμα της Επιτροπής. Για τις τροπολογίες είχε υπάρξει προθεσμία μέχρι τις 12 Αυγούστου και μέχρι τις 25 για όλες τις ε, γλώσσες και για γαλλικά αγγλικά μέχρι τις 25 Αυγούστου. Ο συντάκτης ήταν και είναι ο κύριος Στάσνη. Πίτερ θα θέλατε να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε όπως είπατε. Δεν ήταν πολυβολικές οι προθεσμίες, εν πάση περιπτώσει χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία τα καταφέραμε, παρότι ήμασταν σε διακοπές. Και είμαι ικανοποιημένο γιατί είναι σημαντικό ορισμένα πράγματα να μην καθυστερούν. Για το τμήμα της Κομισιόν θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δύο ήταν οι σημαντικές ανησυχίες της ΙΝΤΑ για τον προπολογισμό της Κομισιόν. Πρώτο, επαρκής χρηματοδότηση για τους τομείς που είναι της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας και δεύτερο, η ίντα να έχει έγκαιρα λεπτομερείς πληροφορίες για την χρηματοδότηση αυτή, που αφενός είναι σημαντική για να μπορούμε να αξιολογήσουμε εάν είναι επαρκές το επίπεδο χρηματοδότησης και από την άλλη για να μπορούμε να παρακολουθούμε την χρηματοδότηση. Οι ανησυχίες που μας απασχόλησαν λοιπόν ήταν αυτές και σας παρακαλώ να με υποστηρίξετε. Θα ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους για την ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία μέσω των τροπολογιών. Και υποστηρίζω την τροπολογία του κυρίου Μάρτιν 6801. Αυτά είναι τα σχόλιά μου για το τμήμα της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Πίτερ. Άλλος κανείς δεν ζητεί το λόγο. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 6804. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ένα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Δύο τροπολογίες τώρα, 6802 ε, και 03, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές απορρίπτεται ή απορρίπτονται. 68.05 και 07. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Μόνο 68.05. 68.05. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6807. Α, αυτή εδώ εκπίπτει. 6808 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6809. Εκπίπτει τελική ψηφοφορία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Χρειάζεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όχι, απαντά ο γραμματέας. Τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2010. Μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν έχετε σχόλια, πείτε Αν ναι, θέλετε να πείτε κάτι. Πολύ σύντομα. Σύντομη εισαγωγή, ώστε οι συναδελφοί μου να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει δυνατότητα για την ίντα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου για, τις, για τους εξωτερικούς τομείς και για τον ΠΟΕ, αντιπροσωπείες, ε, διασκέψεις κοινοβουλευτικών οργάνων κλπ. το σχέδιο γνωμοδότησής μου έχει τρεις στόχους. Πρώτο, να τονίσει και να εξηγήσει τις δραστηριότητες που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ. Πρώτες τρεις παράγραφοι αυτό. Δεύτερο, να σημειώσει ότι θα υπάρχει συνεχώς στο μέλλον η ανάγκη χρηματοδότησης αυτής της ε, δραστηριότητας. Για το 2010 θα γίνει τουλάχιστον μία ε, συνάντηση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΠΟΕ, είτε εκ παραλίλου με τις υπουργικές διασκέψεις του ΠΟΕ, θα εξαρτηθεί αυτό από τα αποτελέσματα του γύρου Ντόχα Αλλιώ θα γίνεται στη Βρυξέλλε είτε στη Γενέβη. Και θα γίνει και μια τη steering committee στην Γενέβη. Και όλα αυτά χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση. Άρα χρειάζονται επαρκή πιστώσει που να επιτρέπουν την συμμετοχή με την απαραίτητη υποδομή τη αντιπροσωπεία σε όλε τι συναντήσει, καθώ επίση για την κάλυψη όλων των εξόδων ταξιδίου και παραστάσεων των ε, ε, μέλων των αντιπροσωπιών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ Πίτερ. Ουδέν σχόλιον. Ωραία. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Υπέρ παρακαλώ. Α, ναι, μια στιγμή. Ψηφίζατε παρακαλώ. Πέρασε, όχι ακόμη. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Εσείς δεν έχετε ψηφίσει, Πίτερ. If you go back a, a row, Peter, and just try on the... Right. Okay. Right. Everybody... Ωραία, ψηφίσατε τώρα όλοι. Μια στιγμή παρακαλώ. First one or the second? We're voting on the first amendment. Ah, the first. Number one. Okay, Now, has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες, λοιπόν. Pardon? Well, 18 in favor, 12 against. Nine. Nine. Anybody who didn't vote uh, didn't, doesn't have the voting card. Ποιος άλλος δεν έχει κάρτα. Τέλος πάντων βλέπω 9 υπέρ και 11 κατά. Που σημαίνει ότι απορρίπτεται η ε, τροπολογία. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α ψηφίσουμε το σχέδιο, το σχέδιο γνωμοδοτήσεως. Το σχέδιο εκθέσεω δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλώς προχωρούμε στην τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδοτήσεως και παρακαλώ αυτό θα, αυτή θα ήθελα να γίνει ηλεκτρονικά. είναι για το πρώτο τμήμα της, ε, του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έτος 2010. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Υπέρ 22 και καμία ψήφος κατά. Σας ευχαριστούμε Πίτερ. Right. Can we now move on to item which is the... Το υπαριθμόν 9. Συμφωνίες, οικονομικές συμφωνίες. Όπου πριν από δύο χρόνια είχαν ε, είχαμε συμφωνήσει να αντικαταστήσουμε το καθεστώς των προτιμήσεων με εμπορικές συμφωνίες τις λεγόμενες ΙΠΑ, που είναι συμφωνίες οι οποίες γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χώρες ΑΚΕ και έχουν ως στόχο να άρουν σταδιακά εμπόδια στο εμπόριο σε όλους τους ε, σχετικούς τομείς. Οι διαπραγματεύσεις των νέων συμφωνιών άρχισαν το 2002 με στόχο να μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Επειδή μέχρι τότε θα έλυγε η συμφωνία που ισχύει. Μόνο οι χώρες της Καραϊβικής ξεκίνησαν τέσσερις ε, συμφωνίες ΕΠΑ μέσα στο αρχικά προβλεπόμενο πλαίσιο. Όλες οι άλλες ομάδες χωρών υπέγραψαν ε, προσωρινές συμφωνίες για αγαθά και υπηρεσίες. Από το 2004 η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις με τις διάφορες ομάδες χωρών σε συναντήσεις και κλεισμένων των θυρών, σε συναντήσεις με την Επιτροπή, με πρέσβεις και με φορείς της ε, κοινωνίας των πολιτών. Στις 25 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οκτώ ψηφίσματα, ένα για κάθε μία για κάθε μία από τις συμφωνίες ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Είχαμε βέβαια και μια μακρά μάχη με την Επιτροπή Αναπτύξεως, και αυτό δεν το λένε οι σημειώσει μου, σχετικά με τις αρμοδιότητες των δύο επιτροπών, της δικής μας και ε, της δικής τους. Καταφέραμε να κερδίσουμε τη μάχη, αλλά ήταν μια σκληρή μάχη. Θα θέλαμε να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού βρίσκονται τώρα, πού βρίσκεται τώρα η πρόοδος για την εφαρμογή των ε, συμφωνιών αυτών και ιδίως οι θεσμικές ε, διαρθρώσεις που προβλέπουν. Ο κύριος ή κυρια Παβέτη Ζαμπίλη. Έχετε το λόγο κύριε. Thank you, Chair. Yes, Όπως θα θυμίστε, η συμφωνία υπογράφηκε πέρσι τον Οκτώβριο και προσωρινά εφαρμόζεται από το Δεκέμβριο πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνένεσε νωρίτερα φέτος. Τα Εθνικά Κοινοβούλια και από τις δύο πλευρές ε, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης όπου αυτή απαιτείται. Οι καλυφορο ε, ε, συζητούν πώς θα οργανωθούν για να εφαρμόσουν την συμφωνία, κάτι το οποίο ενέχει αναδιοργάνωση των δομών και συστημάτων σε ό,τι αφορά περιφερειακή οργάνωση των χωρών αυτών, ε, σε σχέση με τις χώρες Καρικόμ και της ε, Δομινικανής Δημοκρατίας για παράδειγμα. Η πρώτη υπουργική διάσκεψη ελπίζουμε να λάβει χώρα το φθινόπωρο. Ολοκληρώνουμε τώρα τις απαραίτητες εργασίες ε, προς προπαρασκευή αυτής της διάσκεψης, κυρίως τους διαδικαστικούς κανόνες. Ε, θα πρέπει να απτυχθούν και τα συστήματα για την υποστήριξη των εργασιών ε, που προχωρούν. Έλαβε χώρα μία συνάντηση τον Ιούλιο επ' αυτού για να καθοριστεί ένα φύλλο πορείας, ένας οδικός χάρτης όπως ε, καμιά φορά λέμε. Ε, έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι εργασίες, η συμφωνία εφαρμόζεται. Τέλος θα ήθελα να υπενθυμίσω τη σημασία του άρθρου 231 της ε, συμφωνίας, ιδιαίτερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι συστήνει μια ε, διακοινοβουλευτική επιτροπή και εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή και οι χώρες Καλιφόρουμ θα πρέπει, θα πρέπει να οργανωθείτε για να δείτε τα της σύστατης αυτού, αυτής της διακοινοβουλευτικής επιτροπής. Πίτερ, Ήμουν εισηγητής για το Καλιφόρουμ Οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η ολοκλήρωση αυτών για τη Γενική ΕΠΑ νομίζω ότι έδειξαν το καλύτερο πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε έντονες εσωτερικές διαφωνίες, ιδεολογικά διστάμενες ε, και αποκλίνουσες απόψεις, αλλά τελικά εξέβραμε συνένεση μεταξύ ημών, κάτι το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με το θεσμικό μας ρόλο. Δώσαμε έτσι σάρκα και οστά στην υπόσχεση που είχαμε δώσει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συσταθεί το Καλιφόρουμ. Το είχαμε υποσχεθεί και το κάναμε. Βεβαίως πρέπει τώρα να παρακολουθούμε τα της εφαρμογής της ΕΠΑ Καλιφόρουμ. δύσκολο έργο, διότι είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη συμφωνία και το είπαμε αυτό και στα πλαίσια των εσωτερικών μας συζητήσεων, πολλά είναι τα άρθρα ανοιχτά σε ερμηνεία όχι προσωπική αλλά τέλο πάντων διαφορετική και νομίζω ότι ρόλος μας σε αυτή την Επιτροπή τα πέντε επόμενα χρόνια όταν έρθει η στιγμή της ε, ενδιάμεσης αναθεώρησης και επαναξιολόγησης να μην μείνουμε στα λόγια αλλά να κάνουμε δουλειά σε βάθος για να είμαστε σίγουροι ότι η αναθεώρηση αυτή θα είναι σωστή και θα γίνει σε βάθος ακόμα και αν χρειαστεί να οδηγήσει σε κατάργηση της ε, ΕΠΑ αυτής, της συμφωνίας αυτής, αν δηλαδή παρελπίδα αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί ως θα επιθυμούσαμε. Αυτό είναι το έργο μας τα επόμενα πέντε χρόνια. Μιλήσαμε με την κοινωνία των πολιτών. Ίσως θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε μια ετήσια συνάντηση με τους εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Θα το δούμε. Πάντως το βασικό στοιχείο, η βασική αν θέλετε επίσημη δομή στην οποία θα κάνουμε αυτές τις αξιολόγησεις είναι η κοινή διακοινοβουλευτική Επιτροπή και εσείς ε, Πρόεδρε προσωπικά πιστώνεστε αυτή την επιτυχία μεταξύ άλλων γιατί ως συντάκτης μιας αρχικότερης γνωμοδότησης που αφορούσε τη γενική μας προσέγγιση έναντι της ΕΠΑ πριν μπούμε δηλαδή της συνολικής συμφωνίας πριν μπούμε στις διάφορες λεπτομέρειες των συγκεκριμένων συμφωνιών είχατε πει ότι θα ήταν απολύτως ευκταίο να συσταθεί μια διακοινοβουλευτική επιτροπή. Έγινε αυτό και πρέπει να δούμε βεβαίως ε, τις λεπτομέρειες, ε, τα της συστάσεως δηλαδή, συμμετοχής, ε, ποια είναι τα μέλη σε την επιτροπή και ούτω καθεξής. Κοίταξα την έκθεση των συντονιστών σήμερα το πρωί, η οποία φαίνεται ότι κινείται πάνω στις ίδιες άδρες γραμμές, δηλαδή ένα μέλος από κάθε μεριά, 15 δηλαδή από μας, 15 από την άλλη πλευρά. Τώρα, αν πούν οι χώρες της Καραϊβικής ότι θέλουν δύο εκπροσώπους για κάθε χώρα, θα πρέπει και εμείς να στείλουμε 30, κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες. Γι' αυτό λέω ένας από εμά και δηλαδή σχέση ένα προς ένα τέλος πάντων. Αυτό εννοώ. 15-15. Τώρα η σύνθεση. Ε, αυτό, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ ποτέ δεν αμφισβήτησα τη σοφία των συντονιστών 10 για μας, 4 για την Επιτροπή Ανάπτυξης προτείνεται, είναι ένας λογικός συμβιβασμός. 14, 15, τέλο πάντων, 9, 6, ανάλογα με το αν θα είναι 14 ή 15, αν θα έρθει ο Χάρτλι ή όχι. Πάντως είναι κυρίως εμπορικό θέμα, άρα εμείς θα πρέπει να έχουμε την πρωτοκαθεδρία, ίσως ό,τι αφορά την εκπροσώπηση. Λοιπόν, αυτέ οι συναντήσεις θα είναι πολύ σημαντικές τη κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινοβουλευτική, να το πω έτσι, θεώρηση των πραγμάτων και όχι γραφειοκρατική ή κυβερνητική αμυγός. Είναι σημαντικό λοιπόν να παρακολουθούμε τακτικά τις συζητήσεις που θα γίνονται τα επόμενα πέντε χρόνια και νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε σε ποιο ακριβώς σημείο θα λάβει χώρα η πενταετής ενδιάμεση επαναξιολόγηση. Δηλαδή από πότε θα μετρήσουμε τη μεταετή περίοδο από τη θέση ισχύ, από την υπογραφή, από την ε, επικύρωση. Από την υπογραφή εγώ πιστεύω, τον Οκτώβριο δηλαδή. του Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η επαναξιολόγηση θα γίνει τον Οκτώβριο του 2013. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κοίταξε, νομίζω ότι το Καλιφόρουμ θα αποτελέσει ούτως ή Ευχαριστώ Επιτροπή επιθυμεί να ομιλήσει εκ νέου. Όχι. Λοιπόν, David, να σε ευχαριστήσω εκ νέου για τη δουλειά σου. Όσοι συμμετείχαν ε, στο, στην προσπάθεια αυτή, και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, ε, δούλεψαν πολύ σκληρά και νομίζω ότι θα πρέπει να συγχαρούμε την Επιτροπή αυτή για το πώς ε, διεύθυνε τις εργασίες αυτές. Αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα παράδειγμα, ένα προηγούμενο που θα πρέπει να μας κάνει περήφανος. Σας ευχαριστώ λοιπόν εκ νέου. Καλώς. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια... Thank Ας περάσουμε τώρα στην παρουσίαση σχετικά με την ειδική αντιπροσωπεία στο εργαστήριο για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης που διοργάνωσε στην Αντίσα Μπέμπα η Επιτροπή Αφρικανικής Ένωσης. <clears throat> Αναφέρθηκε α, ήδη ότι από το 2004 ε, η Επιτροπή μας ε, παρακολουθεί αυτές τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης Υπάρχει ένα μέλο εκεί, αλλά δεν είναι παρόν. Όχι, είναι παρόν. Δεν σα είχα δει. Συγγνώμη. Ήσασταν μέλος, ε, συμμετείχατε μάλλον σε εργασίες του εργαστηρίου για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης στην Αντίσα Μπέμπα. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ και θα ακούσουμε με ενδιαφέρον όλα όσα έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν δεν έχετε αντίληψη, θα μιλήσω ισπανικά. Όντως είχα την ε, τιμή να εκπροσωπήσω την Επιτροπή μας ε, αλλά και το Κοινοβούλιο διότι κανείς άλλος δεν είχε τη δυνατότητα να παραστεί, λογικό λόγω των ε, εκλογών. Πήγα λοιπόν στην Αντίσα 29 και 30 Ιουλίου όπως ξέρετε, είναι η πρωτεύουσα της Αφρικανικής Ένωσης. Είχαμε λοιπόν μια συνάντηση ακριβώς για το θέμα αυτό, τον ΕΠΑ δηλαδή. Συνάντηση ε, στην οποία παρέστησαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι διαφόρων Αφρικανικών Κοινοβουλίων, εκπρόσωποι του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, αλλά και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Ε, όσο δυνατόν πιο σύντομα θα σας περιγράψω το περιεχόμενο των ε, διαμυφθησών εργασιών. Ήταν τιμή μου που εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπα και προηγουμένως, και ως νέο μέλος και πήγα με ταπεινοφροσύνη λοιπόν και με τριοπάθεια να μιλήσω για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω και απ' έξω και ανακατοτά. Με τη βοήθεια βεβαίως της γραμματείας, ε, χάρη στην οποία μπόρεσα να μάθω πολλά, πήγαν τα πράγματα κατευχήν. Ήθελα να το πω και αυτό. Έκανα μια παρουσίαση του θέματος των ΕΠΑ και επειδή είναι τώρα πρόεδρος ε, ο κύριος Στέρντι, έτσι αισθάνομαι κάπως αμήχανος ε, που θα του απονείμω τα εύσημα, αλλά το γνωρίζετε όλοι ότι έχει κάνει μεγάλη δουλειά ο κύριος Στέρντι επί του θέματος αυτού, το άκουσα και επί τόπου. Επίσης, πολύ θετική ήταν η αντίδραση εκ μέρους της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης και των εκεί περισταμένων για το γεγονός ότι ε, ένας εκπρόσωπος ε, της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, ο υποφαινόμενος στην περίπτωση αυτή, ε, παρουσιάστηκε κάποια στιγμή, εμφανίστηκε με σάρκα και ωστά και αυτό αποτέλεσε ευτυχές γεγονός για όλους. Ο ρόλος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό τον έπαιρνε πολύ σημαντικό, τώρα που συζητούμε τα της εφαρμογή αυτών και η μέρημνα, η ανησυχία αν θέλετε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να ε, μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και να διευκολύνουμε την διαδικασία ολοκλήρωσης ε, της αφρικανικής οικονομίας μεταξύ των διαφορετικών χωρών και την ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία. Προφανώς υποστηρίζουμε πάντα την σωστή και βιώσιμη μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης που θα πρέπει να λάβει η χώρα στις χώρες αυτές. Με τα οκτώ ψηφίσματα του Μαρτίου που και εσείς κύριε Στέρντι αναφέρατε, υπενθύμησα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα παρόν σε τέτοιου είδου διαπραγματεύσει και ανέφερα, υπογράμμισα την σημασία του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια ας πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε τακτικές επαφές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά, κάτι το οποίο έγινε. Υπενθύμησα ότι αυτό το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή είχε ζητήσει την σύσταση μικτών κοινοβουλευτικών δηλαδή συναντήσεων μεταξύ της Επιτροπής μας και των εκπροσώπων των περιφερειών και περιοχών που διαπραγματεύονται είναι δηλαδή υπεύθυνε για τη διαπραγματεύση των ΕΠΑ. Εις ό,τι αφορά τη συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών, τα μέλη των διαφορετικών Αφρικανικών κοινοβουλίων και τα μέλη του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να πω ότι κοινό σημείο ήταν ε, στις παρεμβάσεις όλων η συμμετοχή, ε, η σωστή και δυνατή ισχυρή συμμετοχή της, οργανωνίας των, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, κάτι το οποίο ισχύει, το υπογράμμισαν όλοι, υπάρχουν πολλά think tanks, δεξαμενές σκέψεως δηλαδή, που λειτουργούν θετικά. Ε, κάποια επίκριση ασκήθηκε εναντί του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ΕΠΑ. Δηλαδή ε, το σκιάχτρο του κυρίου Μάντελσον ε, αναφέρθηκε. Όχι ονομαστικά, αλλά μου είπαν α πούμε ότι κοιτάξτε εμεί δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον κύριο Μάντελσον κάτι το οποίο στην αγγλική We are not in love with Mr. Mandelson αποτελεί έναν ε, ένα σχήμα λιτότητος που ουσιαστικά σημαίνει το αντίθετο τέλος απάντων έγινε και μια πρόταση που θεώρησα ευτυχή να έχουμε τακτικές συναντήσεις μεταξύ των δικών μας εκπροσώπων και της ε, Αρμόδιας Επιτροπής της Παναφρικανικής Ένωσης ε, για τα τελωνία και τις ε, εμπορικέ ε, ροέ. Για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, τη ΕΠΑ δηλαδή και άλλα κοινά, κοινού θέματα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα ολοκληρώνοντα να πω το εξής. Εκ μέρους της αφρικανικής πλευράς ε, υπήρξε έντονη και πάγια επιμονή επί του ότι η ΕΠΑ θα πρέπει να βοηθήσουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης και ένταξης ε, της αφρικανικής οικονομίας στην παγκόσμια σκηνή και ότι θα πρέπει να αποτελέσουν ένα μέσο, η ΕΠΑ δηλαδή, βιώσιμης βοήθειας και υποστήριξης αυτής της δικασίας. Προτάσεις. Σας διαβάζω και παραθέτω κατά λέξη. Τα εθνικά και περιφερειακά αφρικανικά κοινοβούλια θα πρέπει να ασκήσουν το έργο της παρακολούθησης monitoring για την εφαρμογή των ΕΠΑ και να παρακολουθούν εκ του στη διαδικασία συζήτησης, διαμόρφωσης και εκτέλεσης ε, εφαρμογής δηλαδή των συγκεκριμένων ΕΠΑ. Με άλλα λόγια, η αφρικανική πλευρά ε, ανέφερε ότι τα Αφρικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν ένα ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη προτάθηκε η σύσταση ενός περιφερειακού φόρουμ και μιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των κοινοβουλίων, των διεθνών οργανώσεων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών με στόχο την προώθηση μιας δημόσιας συμμετοχής, μιας συμμετοχής δηλαδή του πολίτη και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Και τρίτον, προτάθηκε επισήμως η σύσταση κοινών, μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, διακοινοβουλευτικών επιτροπών δηλαδή, όπως λέγαμε και προηγουμένως, για την εξέταση των θεμάτων που εμπίπτουν ε, στο ενδιαφέρον μας. Και αυτές οι διακοινοβουλευτικές επιτροπές ε, θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να υποβάλουν προτάσεις σε σχέση με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω κάτι που είπα και στην αρχή, ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συμμετοχή μου στις εργασίες αυτές. Ε, όπως είπα και προηγουμένως και οι ίδιοι Αφρικανοί εκπρόσωποι ε, εκτίμησαν την ε, παρουσία μου στην Αντίσα Δεδομένων όλων αυτών λοιπόν των στοιχείων και θετικών ενδείξεων πιστεύω ότι ήταν σημαντική πολιτική με την ευρία έννοια του όρου πράξη, κάτι το οποίο εκτιμήθηκε και κάτι το οποίο τονίζει και αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Είσαστε νέος σε αυτή την Επιτροπή και είσαστε νέος ε, στις, ε, στην παρατήρηση αυτή των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και όμως μας ε, εντυπωσιάσατε με τις γνώσεις σας. και μπορούμε να πούμε νομίζω ότι με την αλλαγή του Επιτρόπου άλλαξε και η θέση η στάση της Επιτροπής και μάλλον προς το καλύτερο. Το είπα και εγώ αυτό στην Αδίσα Μπέπα. Ε, το είπα με πολύ ήπιο και λεπτό και διπλωματικό τρόπο, αλλά το είπα πάντως. Ότι τα, πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Ίσως εγώ δεν είμαι τόσο διπλωμάτης και τόσο λεπτό στις εκφράσεις μου. Έχουμε ή έχετε σχόλια, παρατηρήσεις. Ο κ. Σαρίφ. Ευχαριστώ τον Εμίλιο για την ακρίβεια της παρουσίασής του και την εκπροσώπησή μας. Σε αυτά που μας είπε βρίσκουμε κάποιες από τις ανησυχίες που είχαμε υπογραμμίσει ε, στις εκθέσεις μας για την Αφρικανική Ένωση. Η θέση των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι μία από αυτές τις ανησυχίες. Ε, διότι ακούστηκαν διάφορες φωνές ότι ίσως ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων να μην, είναι, πρέπει, δεν πρέπει να είναι τόσο σημαντικός. Αλλά αυτό τονίστηκε. Ε, μια άλλη ανησυχία ήταν η περιφερειακή ολοκλήρωση σε διάφορες ε, διαπραγματεύσεις που κάνουμε με διάφορες ε, χώρες, βλέπουμε ότι ε, έχει αποτύχει αυτή η περιφερειακή ολοκλήρωση. Ενώ αυτή βρισκόταν στον πυρήνα των συμφωνιών. Τρίτον, προσοχή θα πρέπει να δώσουμε και εμείς, αλλά φαίνεται και στους Αφρικανούς εταίρους μας αυτή η ανησυχία, ότι συχνά υπάρχει μία έλλειψη σεβασμού προς τα συμφέροντα των Αφρικανών εταίρων, ειδικά για το θέμα της Σιγκαπούρης. Δηλαδή, τι πίεση ασκούμε στους Αφρικανούς σε σχέση με άλλες χώρες. Για να βοηθήσουν αυτές οι συμφωνίες στην ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε πώς γίνονται και οι διαπραγματεύσεις και πώς αντιμετωπίζουμε τις αφρικανικές χώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Άλλα σχόλια. Η Κομισιόν θέλει να σχολιάσει. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πρόεδρε, δεν έφτασε ακόμα. Θα έρθει σε λίγο όμως. Well, um, I have to say that it was on the agenda. Uh, το ήξερε. ήταν στη μερίσια διάταξη αυτό το σημείο των ε, Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Μάλλον βγήκε, έφυγε δηλαδή, αλλά καλό, καλό θα ήταν να έχει μείνει στην αίθουσα να τελειώσουμε τη συζήτηση. Το επόμενο σημείο θα είναι η παρουσίαση του Κινέζου πρέσβη. Ε, ο πρέσβης αυτός θα έρθει με τον διερμηνέα του. Ίσως λοιπόν να υπάρχει, να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Τον περιμένουμε στις 10 η ώρα. Αν λοιπόν δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο για τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, μπορούμε να σταματήσουμε. Θα ήθελα λίγο να επανέλθουμε στο προηγούμενο σημείο για λίγα λεφτά, γιατί κάτι ξέχασα να πω. Και καλό είναι να το πούμε. Παρότι η Επιτροπή Παρακολούθησης για τις ε, συμφωνίες αυτές ε, στο Καριφόρουμ είναι αυτοτελείς ε, επιτροπές, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνεργάζονται με την μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση. Θα πρέπει δηλαδή να συντονιζόμαστε ως προς τις ε, συνεδριάσεις μας και να μην γίνεται επικάλυψη των ε, προσπαθειών. Γιατί υπάρχουν θέματα πόρων ε, για την Καρεβική, για το, την προσέλευση και την παρουσία στις ε, επιτροπές. Επομένως έχει νόημα να δούμε, να συντονιστούμε. Σίγουρα θα συνεργαστούμε με τις χώρες ΑΚΕ. Δεν έχει νόημα να έχουμε συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης χωρίς συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ. Αλλά καλά έκανες και το έθεσε αυτό το θέμα της, του συντονισμού και της συνεργασίας. Άλλα σχόλια. Ευχαριστώ και κύριε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μέντες Ντεβάγε. Ε, σίγουρα οι γνώση σας για τις εξωτερικές υποθέσεις σας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή την, ε, την περίπτωση. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο αρμόδιος για το θέμα της Αντισαμπέμπα, μόλις έφτασε. Would he Να σχολιάσετε, αλλά σύντομα παρακαλώ. Διότι σε λίγα λεπτά θα φτάσει ο Κινέζος πρέσβης. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Δύο σχόλια. Έχουμε μια στρατηγική με την Αφρικανική Ένωση, η οποία ε, συμπεριλαμβάνει και τη συνεργασία, την εταιρική σχέση ε, για, το περιφερειακό εμπόριο και το διάλογο. Και γι' αυτό λοιπόν συζητάμε με τις χώρες αυτές για τα TBT, για τα τεχνικά, τους τεχνικούς φραγμούς, ε, τα προβλήματα των Αφρικανών με τις εξαγωγές, λόγω έλλειψης του δυναμικού να σεβαστούν τα πρότυπα. Αυτό προωθούμε στη σχέση μας με την Αφρικανική Ένωση και σε στενές επαφές ε, στα πλαίσια των ε, Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, όπου, έχουμε, όπου παίζουμε ένα συντονιστικό ρόλο με, τις, ε, με διάφορες ομάδες αφρικανικών χωρών. Φυσικά όλα αυτά τα θέματα συζητώνται πολύ έντονα. Έχουμε την τη ρήτρα προσαρμογής. Ανάλογα με τον τομέα υπάρχει διαφορετική συμμετοχή. Και αφού υπογράφουμε με τις χώρες και τις ε, περιφέρειες, έχουμε πρωτοβουλίες ε, βοήθειας για το εμπόριο και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να θα βοηθήσουμε να ξεπεράσουν οποιαδήποτε προβλήματα έχουν. David, θες να σχολιάσεις, κύριε Αρίφ? Όχι. Πολύ ωραία. Και τώρα θα περιμένουμε τον Κινέζο πρέσβη. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Θα ζητήσω πρώτα από την Κομισιόν να μιλήσει. Ε, δεν θέλω να δείξω ασέβεια προς τον πρέσβη, αλλά είναι μια νέα επιτροπή αυτή και θα ήθελα να μας θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και εν συνεχεία ο πρέσβης θα σχολιάσει. Καλωσορίζω τον πρέσβη, ο οποίος κάθεται στο βάθος της αίθουσα, Σαν Ζέι, ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομα. Ακούσαμε χθε ότι η Κίνα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, δεύτερος για την, ε, Ευρωπαϊκή, για την, ε, για τη ΣΥΠΑ, συγγνώμη. Όσοι από εσά είχατε παραστεί στο Χονγκ Κόνγκ, στο γύρο της Ντόχα, όπου ήταν παρόντες και οι Κινέζοι, θα θυμάστε ότι η Υπουργοί Εμπορίου ήταν ε, παρόντες ε, μαζί με τους Κινέζους ομολόγους τους. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας ε, θέσει το πλαίσιο. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για ένα πρόβλημα συντονισμού που είχαμε ίσως να οφείλεται στο ότι είναι νέα η Επιτροπή αυτή και ότι ετοιμάζουμε κάποια δελτία, τεχνικά δελτία, για τα πολυάριθμα θέματα τα οποία θα εξετάσετε στην Επιτροπή σας. Γι' αυτό λοιπόν ε, είχαμε εστιάσει περισσότερο στα τεχνικά δελτία και ξεχάσαμε λιγάκι το θέμα του συντονισμού, γι' αυτό χρειάστηκε να περιμένετε. Θα, θα δώσω το λόγο κατευθείαν στο συνάδελφό μου να μιλήσει για την Κίνα. Στη συνάδελφό μου. Όπως αναφέρθηκε ήδη από τον πρόεδρο, οι εμπορικές μας σχέσεις ε, με την Κίνα είναι από τις πιο σημαντικές εμπορικές σχέσεις που έχουμε. Είναι ο δεύτερος ε, ε, εμπορικός εταίρος μετά της ΕΠΑ και είναι μια εμπορική σχέση εύρωστη. Η συνεργασία, η συνεργασία όπως θα ακούσατε, χθες στην Επιτροπή είναι στον πυρήνα της σχέσης, αλλά προφανώς με ένα τέτοιο εμπορικό εταίρο έχουμε και τριβές. Είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εμπορικές σχέσεις, όχι μόνο λόγω του μεγέθους των εμπορικών ροών, αλλά υπάρχουν, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές εμπορικές. Η Κίνα είναι ένας ε, σχετικά νέος εταίρος των ΠΟΕ, στο διεθνές εμπόριο. Την τελευταία δεκαετία είχε μια θεαματική ανάπτυξη, αλλά μαζί με αυτό τα συμπαρομαρτούντα είναι και κάποιες εντάσεις, κάποιες τριβές και η Κίνα χρησιμοποιεί και το βάρος της αυτό ασκεί μια πίεση στις εμπορικές σχέσεις. Ε, θα έχετε ακούσει ότι υπάρχει ένα σημαντικό εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα. 270 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, περίπου. Οι εμπορικές σχέσεις πάντα εμπεριέχουν και διαφορές ε, όταν υπάρχουν πλεονάσματα από τη μία πλευρά και ελλείμματα. το έλλειμμα απέναντι στην Κίνα ή το πλεόνασμα της Κίνας απέναντι μόνο δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο συστημικό πρόβλημα. Αλλά το μέγεθο ε, του ελλείμματο μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικέ εντάσει σε ορισμένε χώρε. Γιατί κάποιε βιομηχανίε ε, επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την ανάπτυξη του εμπορίου τη Κίνα από ότι κάποιε άλλε χώρε. Έχουν γίνει συζητήσει για το εμπορικό έλλειμμα και το αν θα μειωθεί φέτο ή όχι. Αλλά είναι πολύ νωρί για να προβλέψουμε κάτι τέτοιο. Ε, το οικονομικό και εμπορικό κλίμα ε, πέρυσι ήταν πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο και μάλλον θα συνεχιστεί έτσι. Έχει υπάρξει μία μείωση κατά 8% τους πρώτους ε, πέντε μήνες. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση ή αν ε, ανακάμψει το δεύτερο εξάμεινο η οικονομία, μπορεί να μειωθεί κάπως το έλλειμμα, αλλά όχι θεαματικά. Η Κίνα είναι η κινα ειναι μια πολύ σημαντική αγορά για τις ε, ευρωπαϊκές εξαγωγές. Παρότι οι δικές μας εξαγωγές σε σύγκριση με τις εξαγωγές της Κίνας προς εμάς είναι μάλλον μικρές είναι 78 δισεκατομμύρια το 2008 σε σχέση με τα 250 προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι μια αγορά που έχει μια αυξανόμενη μεσαία τάξη, όπου τα ευρωπαϊκά προϊόντα μπορεί να είναι ανταγωνιστικά. Ε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θέλουν και να επενδύσουν και να κάνουν εμπόριο με την Κίνα Τώρα, από την κινέζικη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η νούμερο ένα αγορά εξαγωγών πάνω από την Αμερικανική αγορά. Ε, είμαστε και η μεγαλύτερη πηγή ε, τεχνολογίας πάνω από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Η Κίνα έγινε μέλος στον ΠΟΕ, το είπα και προηγουμένως, έγινε το 2001. Όταν εντάχθηκε στο 2001, ε, ανέλαβε κάποιες δεσμεύσεις για τους δασμούς και μία βαθμία απελευθέρωση άλλων τομέων. Εμείς ε, θέλαμε τότε να μπει η Κίνα στον ΠΟΕ, να γίνει τμήμα του διεθνούς εμπορικού κλίματος και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πιστεύαμε τότε και το πιστεύουμε ακόμα, ε, θα κέρδιζαν και η ΜΕΝ και η ΔΕ. Και τα μέλη του ΠΟΕ και η Κίνα. Φυσικά το εμπόριο ε, ήταν ο πυρήνας και η βασική αιτία της ανάπτυξης της Κίνας τελευταία δεκαετία. Ας περάσουμε στον τομέα των επιχειρήσεων. Πώς ε, κάνουμε ε, πώς αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις μας. Υπάρχουν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στην Κίνα. Αλλάζουν οι τομείς που αναπτύσσονται, αλλά η τάση είναι να γίνονται περισσότερες επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία στην Κίνα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν στην Κίνα επενδύουν για να εξάγουν, όχι για να επανεξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να πουλήσουν στην κινέζικη αγορά. Υπάρχει μια οργάνωση εμπορική εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και επίσης ένα επιμελητήριο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Ε, Κάθε χρόνο αυτά, αυτές οι οργανώσεις συγκρίνουν τι ακριβώς συνέβη, ε, ποιες είναι δυσκολίες ε, και δίνουν συμβουλές στις κινέζικες αρχές για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί το κλίμα. Τον Ιούνιο έγινε μια έρευνα, τον Ιούνιο του 2009, και κάποιες από τις πτυχές της έρευνας αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, λέει η έρευνα, που δραστηριοποιούνται στην Κίνα λένε ότι επηρεάστηκαν από την κρίση, ίσως λόγω της μείωσης της εσωτερικής, της εγχώριας κατανάλωσης. Πάνω από το 70% των επιχειρήσεων είπαν ότι η κινέζικη αγορά ήταν πιο ανθεκτική στην κρίση από άλλες αγορές, ακόμα και από την ε, ευρωπαϊκή αγορά. 50% και παραπάνω πιστεύουν, από τις επιχειρήσεις, πιστεύουν ότι η κρίση στην Κίνα θα τελειώσει μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2010. Το μέλλον δηλαδή προβλέπεται καλύτερο για την Κίνα. Για το πακέτο ενθάρρυνσης. 10% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετό για να κρατήσει την οικονομική ανάπτυξη το 2009. Επίσης, 50% των επιχειρήσεων ε, πιστεύουν ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη αν υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, ο οποίος θα σπάσει τα μονοπόλια. Επίσης, ε, το Κινέζικο Εμπορικό Επιμελητήριο έρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ε, να επισκεφθεί την Ευρώπη, το, τους ομόλογούς τους. Συνήθως η επίσκεψη γίνεται το Σεπτέμβριο για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2006 ε, εκδόθηκε μία ανακοίνωση που είναι η βάση για τη συνεργασία ε, με την Κίνα. Υπάρχει ένα κείμενο επίσης ε, για την εταιρική σχέση και τη συνεργασία με την Κίνα. Σε αυτό το έγγραφο ε, τίθεται το πλαίσιο για τη συνεργασία και την εμπορική, και την εμπορική εταιρική σχέση. Επίσης συζητήσαμε για το τι γίνεται όταν η συνεργασία και ο διάλογος δεν προχωρούν. Η βασική αρχή είναι σαφής, ότι αξιολογούμε τις δεσμεύσεις της Κίνας προ... απέναντι στον ΠΟΕ, βλέπουμε πού υπάρχουν κενά και αν κάποιες δυσκολίες δεν μπορούν να επιληθούν, κοιτάμε άλλες εναλλακτικέ λύσεις, όπως κάνουμε και εμάς τους εμπορικούς εταίρους. Αν θα προσφύγουμε σε πάνελ του ΠΟΕ, όπως έχουμε κάνει τρεις φορές τα περασμένα χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούμε να διορθώσουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν όμως ε, στενές επαφές με τις κινέζικες ε, αρχές και με τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης, μία φορά το χρόνο υπάρχει μία σύνδοση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και τα εμπορικά θέματα είναι πολύ ψηλά στη μερισία διάταξη. Ίσως να θυμάστε ότι η σύνδοση κορυφής το 2008 αναβλήθηκε και, θα γίνει, και έγινε το πρώτο μισό του 2009 και η δεύτερη σύνοδος θα γίνει και αυτή μέσα στο 2009. Ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένη για το 2009. Έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο διαλόγου για οικονομικά και εμπορικά θέματα. η Επίτροπος Άστον είναι επικεφαλής αυτής της Επιτροπής που ασχολείται με αυτά τα θέματα και αυτός ο διάλογος υψηλού επίπεδου για οικονομικά και εμπορικά θέματα ε, συστήθηκε για να εξεταστούν διάφορα θέματα για το εμπόριο και τις επενδύσεις που δεν εντάσσονται στο, στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορίου ε, στην Κίνα. Ε, δηλαδή εκεί που εμπλέκονται διαφορετικά υπουργεία στην Κίνα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τέτοιου τύπου ε, κανάλια για να μπορούμε να επηρεάσουμε το ε, εμπόριο και τις επενδύσεις. Το εμπόριο και οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν. και αυτή η επιτροπή είναι πιο στρατηγική από άλλες επιτροπές που έχουμε. Έχουμε μία μεικτή επιτροπή επίσης που τη συμπροεδρεύει ο, εμπορ, ο Επίτροπος Εμπορίου και Εξωτερικών Σχέσεων και εκεί ασχολούμαστε περισσότερο με εμπορικά θέματα. Συζητάμε την τεχνική αρρωγή επίσης, ε, εξού και η συμμετοχή από τη ΡΕΛΕΞ. Και κάτω από αυτό το επίπεδο έχουμε διάφορες επιτροπές, ε, ομάδες εργασίας, ε, σε επίπεδο γενικών διευθυντών, σε επίπεδο διευθυντών, σε επίπεδο τμήματαρχών ακόμα. Επίσης έχουμε ομάδες εργασίας για συγκεκριμένα θέματα όπως ε, κρυστοφαντουργικά, χάλιβας, ε, αηφόρος ανάπτυξη. Προτιμούμε το διάλογο, όπως σας είπα, για τις εργασίες μας. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένε περιπτώσεις, χρειάστηκε να προσφύγουμε στην, στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μία φορά για τις εισαγωγές αυτοκινήτων, ε, για τα συγγνώμη, εξαρτήματα αυτοκινήτων, για την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και μία τρίτη για τις πρώτες σύγκλες. Τρίτη προσφυγή. Κάτι άλλο που ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο είναι οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες συνεργασίας και εταιρικής σχέσης. Αυτές οι συμφωνίες Αυτές οι διαπραγματεύσεις μάλλον επίσημα ξεκίνησαν το 2007 και προχωρούμε παράλληλα σε δύο τραπούς. Έχουμε το πολιτικό στοιχείο ε, με τον Επίτροπο Εξωτερικών Υποθέσεων και έχουμε τον, την εμπορική, τα εμπορικά θέματα. Τα τελευταία δύο χρόνια διαπραγματευόμαστε και από ευρωπαϊκής πλευράς θέλουμε να υπάρξει μια φιλόδοξη συμφωνία που θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες ε, δεκαετίες για την ε, βιομηχανία μας, ε, για το εμπόριο με την Κίνα. Δυστυχώς καθυστέρησαν λίγο οι διαπραγματεύσεις για τα εμπορικά θέματα, φυσικά είναι περίπλοκες και είναι πολύ σημαντικές για τη βιομηχανία ένθεν και ένθεν. Πιστεύουμε παρόλα αυτά ότι θα επιταχυνθούν την άνοιξη που μας έρχεται και θα συμφωνήσουμε σε κάποια άρθρα μέχρι να φτάσουμε στη συνοκορυφή. Για τα εμπορικά θέματα, αυτέ οι συμφωνίε δεν είναι ελευθέρου εμπορίου, έτσι. Επομένω, δεν διαπραγματευόμαστε δασμού. Η απόφαση ελήφθη πριν τη διαπραγματεύση να μην μπούμε στα θέματα των δασμών. Οι δασμοί της Κίνας μετά την προσχώρηση της ε, Κίνας ε, στον ΠΟΕ είναι σχετικά ε, χαμηλή, είναι κάτω από το 10%. Ίσως θα ήταν υπερβολικά φιλόδοξο να υπησέλθουμε σε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις ξανά. Εξάλλου υπάρχουν και κάποιες δικές μας ευαισθησίες για τα θέματα αυτά. Για τις επενδύσεις, αυτό είναι, μια, αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για τη συνεργασία μας με την Κίνα. Ελπίζουμε ότι θα προοδεύσουμε τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον τομέα. Μας ενδιαφέρει και εμάς. Έχουμε κάποια κενά επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς ακόμα που συμφωνήθηκαν στον ΠΟΕ, αλλά έχει νόημα να προχωρήσουμε περαιτέρω και από κινέζικης πλευράς υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επενδύουν στην Ευρώπη. Θα θυμάστε τις συζητήσεις για τα κυρίαρχα κρατικά ταμεία που είχαμε πέρυσι επιβεβαιώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή για επενδύσεις σε τέτοιου τύπου ταμεία. Φυσικά συζητάμε το θέμα αυτό, αλλά γενικά είμαστε ανοιχτοί επί της αρχής. Φυσικά θα πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την συνεργασία που ήταν προβληματικό ήταν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις σε αυτό το θέμα, ειδικά για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από παραβιάσεις των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Επίσης, αν δείτε τις στατιστικές των τελωνίων, αν δείτε τα αγωθά τα οποία σταματούμε στα σύνορά μας. Ε, το 54% αυτών ε, στα, τα σταματάμε στα τελωνία γιατί υπάρχουν παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν βελτιώσεις, ειδικά στο νομικό πλαίσιο στην Κίνα, αλλά ακόμα υπάρχουν ελλείψεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σχετικών νόμων και ο διάλογος συνεχίζεται με τις κινέζικες αρχές για το πώς θα υποστηρίξουμε την εφαρμογή των ε, κανόνων και του νομικού συστήματος. Ο Επίτροπος ε, έχει προσπαθήσει να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά, όχι την νομική αρρωγή, αλλά προσπαθεί να εντοπίσει τα κενά, τα προβλήματα και να τα καλύψουμε. Πάμε στην τεχνική αρρωγή. Έχουμε διάφορα προγράμματα και σχέδια τα οποία είναι εξελίξη. Η βασική εστίαση αυτή τη στιγμή είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι η βάση της συνεργασίας μας και συνδέεται με το πρόγραμμα που συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό. Συνδέεται με αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, πώς η Κίνα θα εκπληρώσει τις ε, υποχρεώσεις της απέναντι στον ΠΟΕ. Τον Απρίλιο του 2008 ξεκινήσαμε και όπως σας είπαμε ο σκοπός είναι να δώσουμε συμβουλές στις ε, ευρωπαϊκές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα με τις κινέζικες παραβάσεις. Υπάρχει και ένα κέντρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που άρχισε να λειτουργεί στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο Υπάρχει σχετική χρηματοδότηση που προβλέπεται από τις ε, συμφωνίες εταιρικής ε, σχέσης. Ε, βοηθάμε και με αυτόν τον τρόπο για να εξάγουν οι επιχειρήσεις οι μικρομεσαίες είτε για να επενδύσουν. Και αποτελεί και μια πλατφόρμα για τα ευρωπαϊκά κράτη προκειμένου να υπάρχει συνεργασία για θέματα επενδύσεων. Θα σταματήσω εδώ και ε, μπορώ βεβαίως να απαντήσω αργότερα σε ερωτήσεις, αφού ακούσω πρώτα τον Κινέζο πρέσβη. Ευχαριστώ. Πριν να καλωσορίσω τον πρέσβη, ε, θα ήθελα να θυμίσω ότι έχουμε εγκρίνει ήδη μια σημαντική έκθεση για τις σχέσεις με την Κίνα τον Φεβρουάριο του 2009, νομίζω του κ. Κόουλ, που είχε τονίσει η έκθεση αυτή και ορισμένες από τις ανησυχίες που σημειώνονται, αλλά είχε καταδείξει και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθιξε, οι εκπρόσωπος δηλαδή, πολλά από τα θέματα τα οποία σκεπτόμουν και εγώ. Ορισμένοι θα θυμάστε την νομοθεσία anti-dumping που είχαμε υιοθετήσει και που είχε, ε, ήταν κάπως μια τραυματική εμπειρία και για την Κίνα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν τέλει. Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί σχέσεις, υπάρχουν μηχανισμοί αντι-dumping κλπ. Είναι σημαντική και για σας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάντως είναι πάντοτε καλύτερος ο διάλογος, άλλωστε λέμε ε, και, ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο κάλιο διαλέγου παρά ε, πόλεμο. Είναι λοιπόν νομίζω αλήθεια ότι οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών επιτρέπουν την ανάπτυξη των οικονομιών όλων των χωρών. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή βέβαια σχεδόν όλε τις οικονομίε του κόσμου να βρίσκονται σε κρίση και για το λόγο αυτό ακόμη είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος. Σας ευχαριστώ για την έλευσή σας σήμερα εδώ και με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τα όσα μας πείτε. Ο πρέσβης, σας ευχαριστώ. Κάποτε ο Πρωθυπουργό σα είχε πει ακριβώ αυτό. Καλύτερα να διαλέγετε κανεί παρά να διεξάγει πόλεμο. <clears throat> Ο Winston Τσόρτσιλ, όπως είπα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που έχω την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας και να συζητήσω θέματα εμπορίου και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της χώρας μου, της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα θα ήθελα να σας συγχαρώ όλες και όλους για την εκλογή σας ως μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας εύχομαι ε, καλή σταδιοδρομία για τα χρόνια που θα ε, βρίσκεστε εδώ. Οι συνάδελφοί μου σας έχουν διανύμει το έγγραφο ε, του λόγου μου, ε, στο οποίο θα ε, βρείτε πολλά στοιχεία και αριθμούς. Επειδή υπάρχει κάποιος περιορισμός χρόνου, θα ήθελα εγώ να περιοριστώ στα πιο σημαντικά θέματα. Όταν εξετάζουμε τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οικονομική και εμπορική συνεργασία, αυτά δηλαδή κυρίως, αυτή, αυτή αναδύεται. Ήδη από το 1975 αρχίσαμε να αναπτύσσουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις και η συνολική μας σχέση έχει συνεχίσει να εξελίσσεται έκτοτε. Γίνεται πιο στέρεα και πιο όρημη, αποφέροντας σημαντικά ωφελήματα στους λαούς μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές ε, στην οικονομική συνεργασία. Θα σας το εξηγήσω, θα σας το εξηγήσω αυτά με βάση τρία θέματα. Πρώτον, έχουμε γίνει πλέον σημαντική εμπορική και οικονομική εταίροι. Σε σύγκριση με το 1975, το εμπόριό μας έχει εξαπλασιαστεί πέρσι και έχει περάσει πλέον και από τα αγαθά και στις υπηρεσίες και στην τεχνολογία. Οι επενδύσεις σας στην Κίνα που ξεκίνησαν σχεδόν από το μηδέν έχουν φτάσει πλέον στα 33,9 δις αμερικανικά δολάρια σήμερα. Οι επενδύσεις της Κίνας επίσης αρχίζουν να έρχονται στην Ευρώπη. Οι επαφές μας για την μεταφορά τεχνολογίας ανέρχεται σε μια αξία 122 δις αμερικανικών δολαρίων. Αυτά τα υψηλά νούμερα εξηγούν και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Κίνας και για εξαγωγές, ως εξαγωγική αγορά δηλαδή, αλλά και ως προμηθευτής τεχνολογίας. Και γιατί η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια εξαγωγική αγορά δυναμικό. Δεύτερο, έχουμε ε, ωφεληθεί τα μέγιστα από αυτή την ε, αμοιβαίως επωφελή συνεργασία. Το χαμηλό κόστος παραγωγής στην Κίνα επιτρέπει στην Ευρώπη να ε, παράγει προϊόντα με πολύ χαμηλότερο κόστος, οδηγώντας έτσι σε μεγάλες εξοικονομήσεις. Παραπάνω από 20.000 ευρωπαϊκές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Κίνα και έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και ε, τα μηχανήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμβάλει σημαντικά στην ε, βιομηχανική αναβάθμιση και οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα παράγουν περισσότερη απασχόληση και έσοδα από φορολογία. Η συνεργασία μας συμβάλλει στην βελτιστοποίηση της, ε, των οικονομικών διαφθρώσεων, αύξηση της παραγωγικότητας και βέβαια της ανάπτυξης. Τρίτο, έχουμε σφυριλατήσει μια στενότερη και σφιχτότερη διμερή συνεργασία. Το εμπόριο και η οικονομική συνεργασία μας κάνουν βεβαίως και πιο εξαρτώμενους. Πολλά αγαθά που κυκλοφορούν σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν ε, παραχθεί στην Κίνα, αλλά και πολλές υπηρεσίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λειτουργούν στην Κίνα. Και ε, παραπάνω από 150.000 Ευρωπαίοι πολίτες εργάζονται στην Κίνα, ενώ παραπάνω από 200.000 ε, Κινέζοι φοιτητέ σπουδάζουν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έχουμε λοιπόν καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεν προς τους δε, το οποίο οδηγεί βεβαίως και στην ε, ανάπτυξη μιας πραγματικής στρατηγικής συνεργασίας. Α, υφίσταται όμως το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στους πρώτους 7 μήνες του έτους το όγκος των συναλλαγών μας ε, μειώθηκε κατά 20 περίπου και οι επενδύσεις κατά, προ, τις δικές σας προς την Κίνα κατά 4,8%. Αποτελεί πραγματική δοκιμασία αυτή η κρίση. Ωστόσο, εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξο για το μέλλον της συνεργασίας μας και για τους εξή τέσσερις λόγους. Πρώτος, στους δύσκολους αυτούς καιρούς η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζονται μια σημαντική συνένεση για να προωθήσουν τους κοινούς στόχους. οικονομική συνεργασία και εμπορική συνεργασία θεωρούμε ότι θα είναι ο μοχλός εκείνος που θα μας επιτρέψει να εξέλθουμε από την κρίση. Σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου και στον οικονομικό και εμπορικό διάλογο οι δύο πλευρές έχουν τονίσει κατά επανάληψη φέτος ότι θα συνεργαστούμε για να καταπολεμήσουμε την κρίση, να προωθήσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις. Αυτά κατεδείχθησαν και με συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τεχνολογιών εχμής και των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Και με σημαντικές παραγγελίες από ε, τις αρχές προμηθειών της Κίνας. Δεύτερο, το πρόγραμμά μας για τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων στις ε, ε, επιχειρήσεις προσφέρει νέες ευκαιρίες. Η κινέζικη κυβέρνηση δραστηριοποιείται στην εφαρμογή ενός προγράμματος παροχής κινήτρων που έχει, ήδη αρχίσει να αποδίδει και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες υπέρ και των αλλοδαπών επιχειρήσεων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι γνωστές για την ε, τεχνολογική τους υπεροχή και, την, ε, ε, και το υψηλό επίπεδο διοικητικής ικανότητας. Και έχουν αποδώσει καλά. Στους πρώτους 7 μήνες οι κινέζικες εισαγωγές από την Ευρώπη μειώθηκαν μόνο κατά 12,2%. Πολύ λιγότερο δηλαδή από, το συνολικό, από τη συνολική μείωση του 23,6%. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες στις προβλέψεις τους προβλέπουν υψηλότερα κέρδη για φέτος και πρόκειται να αυξήσουν τις επενδύσεις τους. Τρίτο, Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σημαντικό δυναμικό αναπτύξεως των αγορών τους. Η Κίνα προσπαθεί να βασίσει και την εσωτερική της ζήτηση και για να γίνει αυτό έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα για να αυξήσουμε το επίπεδο ευημερίας, να βελτιώσουμε την κοινωνική ασφάλεια και να τονώσουμε την ε, ε, ζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι μέχρι το 2010 ο τομέας των, ε, αγαθών υψηλής ποιότητα στην Κίνα θα ανέρχεται στο 1-3 εκατομμύριο δολάρια καταξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη μεριά είναι η σημαντικότερη παγκόσμια καταναλωτική αγορά και ανοίγει σημαντικές ευκαιρίες για τις κινέζικες επιχειρήσεις. Τέταρτο, αλλά και πιο σημαντικό, η Κίνα θα συνεχίσει το άνοιγμά της μέσα σε μια αμοιβαία υποφελή συνεργασία. Αυτή τη στιγμή ενταχθήκαμε στον ΠΟΕ οι γενικοί μας δασμοί κατήθαν από το 15,3% στο 9% περίπου. Έχουμε ανοίξει πολλούς τομείς υπηρεσιών, το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή, και οι εισαγωγές μας ανήλθαν πέρσι στο 1,13 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στο μέλλον η Κίνα θα συνεχίσει να αυξάνει τις εισαγωγές της, κυρίως προηγμένης τεχνολογίας και εξοπλισμού, τμήματων μηχανημάτων, ανταλλακτικών, καθώς επίσης και πρώτων υλών. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις ε, αλλοδαπές επενδύσεις, κυρίως σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ε, σχετικών και συναφών τομέων. Ταυτόχρονα θα ενθαρρύνουμε τις κινέζικες επιχειρήσεις να μεταβούν στην αλλοδαπή διότι θεωρούμε ότι οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν και ε, στην ε, εντόπια απασχόληση. Κυρίε και κύριοι, όπου υπάρχει φως υπάρχουν και σκιές. Υπάρχουν βεβαίως τριβές στις επαφές μας, εμπορικές και επιχειρηματικές. Η κινέζικη πλευρά ανησυχεί για θέματα ε, όπως της αγοράς τροφίμων, όπως ορισμένων περιορισμών ε, στις εξαγωγές και στην ε, χορήγηση προξενικών θεωρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά παραπονιέται για την ανισορροπία του ισοζυγίου συναλλαγών. Αλλά για να ενισχύσουμε τις εμπορικές και οικονομικές μας σχέσεις πρέπει να επιλέξουμε και κάποιες νέες προσεγγίσεις και να δώσουμε μια νέα όθηση. Θα σας κάνω πέντε προτάσεις. Πρώτη, θα τηρήσουμε ή θα, θα παρακολουθήσουμε αν θέλετε τις ε, σχέσεις αυτές και από μακροοικονομική σκοπιά. Έχουμε, ε, έχουν γίνει τόσο στενές οι σχέσεις μας που σίγουρα έχουν και ε, ασκούν επιρροή και σε άλλους τομείς της συνεργασίας μας. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε ορισμένε μεμονωμένες περιπτώσεις να βλάψουν τη συνολική μας συνεργασία. Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας μας για το εμπόριο και για τα οικονομικά θέματα. Μαζί με μια αποτελεσματική άσκηση πολιτικής μέσω διαλόγου. Δεν θα επιτρέψουμε να εκτροχιαστούν αυτές οι προσπάθειες από οποιασδήποτε μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεύτερο, θα τηρήσουμε την αρχή του αμοιβαίου ανοίγματο και της αμοιβαίας ωφέλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε τάχθηκε υπέρ των ανοιχτών αγορών. Η Κίνα επίσης θα τηρήσει την πολιτική του ανοίγματο. Η πολιτική ανοίγματος της Κίνας προσανατολίζεται προς την επιδίωξη μιας κοινή οικονομικής ανάπτυξης. Θα συνεργαστεί η Κίνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διατηρήσει ανοιχτές αγορές και να αποφύγει τον προστατευτισμό. Και θα δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες υπέρ του εμπορίου και των επενδύσεων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν το ε, πλεόνασμα στην Κίνα και λόγω της μεταφοράς επιχειρήσεων στην ε, χώρα μας. Δεν ευθύνεται για το πλεόνασμα αυτό η κινέζικη εμπορική πολιτική. Αντίθετα, η ε, Κίνα έχει κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τονώσει τις εισαγωγέ ακόμα και όταν η κρίση έπληξε τις εξαγωγές μας. Τρίτο, θα διατηρήσουμε και θα βελτιώσουμε τις επικοινωνίες μας και τους μηχανισμούς επαφών. Έχουμε δημιουργήσει έναν μηχανισμό πολυμερή που, στον οποίο συμμετέχουν και ηγετικές προσωπικότητες αλλά και τεχνικό προσωπικό και είναι σημαντικό για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την άρση τους. Τον προηγούμενο Μάιο η ενδέκατη διάσκεψη κορυφής Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δεύτερος διάλογος έπαιξε σημαντικό ρόλο για τη σταθεροποίηση του, των εμπορικών μας σχέσεων μέσα, όπως είπα, σε περίοδο κρίσεως. Στο μέλλον θα κάνουμε καλύτερη χρήση του μηχανισμού αυτού για να διευρύνουμε τις ανταλλαγές απόψεων και σχέσεις και να επιλύουμε τις διαφορές μας. Τέταρτο. Η Κίνα έχει προχωρήσει προς την εκβιομηχάνηση. Η βιομηχανία της γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και θα συνεχίσει να ανθίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη πλευρά είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη οικονομία και η συμμετοχή της σε επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα στην έρευνα και ανάπτυξη παγκόσμια θα συνεχίσει να παραμένει. Αυτός ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των οικονομιών μας ανοίγει ευρύ πεδίο συνεργασίας. Σημαίνει όμως ακόμη ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε πλήρη ισορροπία και στις δύο πλευρές κάθε τομέα. Αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε θα είναι να προσαρμοστούμε καλύτερα, αντί να, να, επιμένουμε στην προστασία των πιο ασθενών α, τομέων μας με τέτοια επιμονή. Τέλος, η παγκόσμια οικονομία περνά από μια σοβαρή κρίση. Όμως θα δώσει, πιστεύω, νέα όθηση στην ε, ανάπτυξη. Η Κίνα επιταχύνει την ε, μεταρρύθμιση του οικονομικού της μοντέλου. Χρειαζόμαστε εμείς εσάς και εσείς εμάς ακόμη περισσότερο. Ακόμα λοιπόν περισσότερη συνεργασία για στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος η συνεργασία μας έχει ήδη επιτύχει κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα σε ορισμένους τομείς όπως της τεχνολογίας εχμής εξακολουθούν να παραμένουν τα προβλήματα λόγω των περιορισμών από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, που ελπίζουμε ότι θα χαλαρώσουν σιγά σιγά. Αξιότιμες κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, ω μέλη τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, είστε τα μέλη της ε, πιο έμπειρης ομάδας ε, προσώπων ε, στον τομέα αυτό. Αντιλαμβανόμαστε τον ενθουσιασμό και τον ζήλο σας για το άνοιγμα των εμπορικών σχέσεων ακόμα περισσότερο με την Κίνα. Και αυτό μας εμπνέει. Ελπίζω θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε περαιτέρω ώστε να δημιουργήσουμε μια θετική ατμόσφαιρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, δημιουργώντας έτσι μια πραγματική στρατηγική σχέση η οποία θα αποβεί αμοιβαία επωφελής για τους λαούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ambassador. I think this is... Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική αρχή που κάνουμε στη νέα μας Επιτροπή, στη νέα μας θητεία δηλαδή, και η παρέμβασή σας ε, καταδεικνύει όχι μόνο ε, τη σημασία που έχει η Επιτροπή μας όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ένωση αλλά και προς τα έξω και ιδιαίτερα στην Κίνα. Προσδοκώ στην αγαστή συνεργασία μας τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο κύκλος ερωταπαντήσεων μπορεί να ξεκινήσει τώρα. ο κύριος Θάλμπα. Στη Σύνοδο Κορυφής, η κυβέρνησή σας και εσείς ο ίδιος είπατε ότι η κινέζικη οικονομία προσαρμόζεται στις παγκόσμιες εξελίξεις. Πώς αυτό συνάδει με τον προστατευτισμό που εφαρμόζεται για τα μη δασμολογικά εμπόδια Προτίθεστε να τα καταργήσετε σταδιακά για να βελτιώσετε τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, ποια είναι η θέση της κυβέρνησής σας για τα φορολογικά κίνητρα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί στην Κινέζικη επικράτεια. Η κυβέρνησή σας προτίθεται να εφαρμόσει τέτοιου είδους φορολογικά κίνητρα ή να τα καταργήσει. Ας απαντηθούν οι ερωτήσεις μία-μία, παρακαλώ. Ζήτω συγγνώμη, αλλά δεν εννοήσα. Θα μπορούσατε να επαναλάβετε. Ο κύριος ε, Στέρντι, καλύτερο θα ήταν να μιλάει ο καθένας τη γλώσσα του. Ο κύριος Θάλμπα, εκ νέου. Ένα λεπτό περιμένετε να βάλει τα ακουστικά το πρέσβης. Στο κανάλι 2 μπορείτε να ακούσετε την αγγλική μετάφραση, λέει στον πρέσβη ο πρόεδρος, ο κύριος Στάλμπα. Ερώτησα, κύριε πρεσβευτά, το εξής. Εφόσον το εμπόριο ε, θα είναι ε, σημαντικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, γιατί η Κίνα προωθεί μέτρα προστατευτισμού με την μη άρση μη δασμολογικών εμποδίων. Προτίθεστε να τα μειώσετε, τα μη δασμολογικά εμπόδια, λόγω της ε, εμπορικής σχέσης που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης θα ήθελα να γνωρίζω τη θέση της ε, κινέζικης κυβέρνησης σε σχέση με τα φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία ξένων επιχειρήσεων, για την εγκατάσταση και δημιουργία ξένων επιχειρήσεων στην Κίνα. Θα άρετε τα μέτρα αυτά. Πρόεδρος, όχι μόνο προς τον κύριο Πρεσβευτή, αλλά και προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορείτε να υπευθύνετε ερωτήματα. Ευχαριστώ. Είμαστε κατά κάθε μορφής προστατευτισμού και δεν δημιουργούμε επουδενή μέτρα διακριτικής μεταχείρισης. Για παράδειγμα, ε, κάποια μέσα ενημέρωσης ε, στο παρελθόν έχουν παρανοήσει τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και υπάρχει μια νομίζω ε, μεροληψία έναντι των μέτρων αυτών. Πρόκειται για παρανόηση, πιστεύω. Τον Ιούνιο φέτος η νέα πολιτική που ισχύει στη χώρα μου είναι υπέρ της νομικής προστασίας των προϊόντων που κατασκευάζονται ε, στην Κίνα συμπεριλαμβανομένου και από ξένες επιχειρήσεις, αλλοδαπές ε, επιχειρήσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να το άνοιγμα των ε, αγορών μας και στον τομέα των δημόσιων προμηθειών και ελπίζω τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια α, ρεαλιστική στάση στα πλαίσια αυτά. Κύριος Ρονάλντι la relazione dell'ambasciatore. Eh, certamente eh, noi siamo tutti molto soddisfatti del grande aumento del volume. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αύξηση του όγκου των εμπορικών ροών μεταξύ ΕΕ και Κίνας και ως ε, ε, φιλελεύθερος ε, πιστεύω ότι ήταν το σημαντικότερο στοιχείο για τη σταθερότητα στον πλανήτη όχι δηλαδή μόνο για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Κίνας. Η σταθερότητα και μια ε, ευημερία παντού είναι οι παράγοντες ε, που θα διασφαλίσουν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, το έλλειμμα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης ε, τα τελευταία χρόνια τριπλασιάστηκε. 50% από το 50% περάσαμε στο 150% ίσως ό,τι αφορά στο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών. Ερώτημα προς τον Πρεσβευτή αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ανάλυση με στοιχεία για το πώς μέσω ή μακροπρόθεσμα διαμορφώνεται η κατάσταση. Είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση του εμπορικού ελλείμματος. Και αυτό βεβαίω άπτεται και άμεσα ε, του θέματος που ανέφερε ο πρεσβής και τον ευχαριστώ για αυτό, της περαιτέρω πρόσβασης των ευρωπαϊκών προϊόντων στην κινέζικη αγορά. Θα ήθελα να γνωρίζω κυρίως εις ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ΕΠΑ που ε, γίνεται με την ε, Κίνα. Και πέραν αυτού, ποιες είναι οι προοπτικές της Κίνας για περαιτέρω άνοιγμα, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, και όπου οι ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα να προσχωρήσουν δηλαδή στην ε, κινέζικη αγορά. Υπάρχει ένα dumping όχι μόνο δασμολογικό αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό και υπάρχει έλλειμμα διαφάνειας ό,τι αφορά την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων, όπως ας πούμε ε, των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιεί ε, ο χημικός τομέας στην Κίνα και που ε, εμείς εισάγουμε για κατασκευή φαρμάκων. Υπάρχει πιστοποίηση υπάρχει, αλλά δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια διαφάνειας και ανιχνευσιμότητα του προϊόντος, όπου εμείς θα θέλαμε. Άλλο πρόβλημα, η αυτοκινητοβιομηχανία, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2009, ε, εξέπνεε η προθεσμία ε, για τον, που είχε λάβει η Κίνα για να σεβαστεί κάποιες υποχρεώσει, υποχρεώσεις της δύναμη του ΠΟΕ. Κάποια ε, ε, κριτήρια, κάποια θέματα που ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε κάποιο πάνελ στον ε, ΠΟΕ, ε, θέματα, προβλήματα με την κινέζικη αυτοβιομηχανία. Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και εδώ ζητώ από τον πρέσβη και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περαιτέρω στοιχεία για αυτή την προσφυγή στο πάνελ του ΠΟΕ. Τώρα, εμείς ως ομάδα, ως πολιτική ομάδα, πάντα θεωρούσαμε ε, την ε, σχέση μας με την Κίνα ως ε, ένα σύνολο που δεν έχει μόνο εμπορικά και οικονομικά θέματα αλλά και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και με τα προβλήματα που έλαβαν χώρα μας ζητήθηκαν πολλές διευκρινήσεις, δεν ξέρω αν έχετε εσείς περισσότερα στοιχεία για τους ανθρώπους αυτούς που αγνοούνται και το σχετικό επεισόδιο. Είναι ένα ερώτημα ρητορικό βεβαίως. Ε, τι γίνεται με τον Λουιτζά ε, που έχει λάβει ε, το βραβείο Ζαχάροφ προβλέπεται αναθεώρηση, προβλέπεται νέα εκδίκαση της ε, υπόθεσης. Θα αποφυλακιστεί. Θέλουμε περισσότερες πληροφορίες από τον πρέσβη. Και ολοκληρώνω με δύο ακόμα ερωτήσεις. Γρήγορα, γρήγορα. Εντάχει Πώς εντάσσεται ε, η χώρα σας ε, στο νότιο, ανατολικό σκηνικό της Ασίας ιδιαίτερα. Αυτό αφορά την Ταϊβάν, τις σχέσεις με την Ταϊβάν, ε, της οποίας η νέα κυβέρνηση πιστεύω ότι ευνοεί εξομάλυνση των σχέσεων. Η επίσκεψή σας στην Ταϊβάν, δεν ξέρω βεβαίως τι συνέπειες θα έχει βαρύες ε, ακόμα και από εμπορική άποψη. Και δεύτερο ερώτημα. Τι πιστεύετε για την αλλαγή κυβέρνηση στην Ιαπωνία. Μετά από 50 χρόνια πέρασε σε άλλα ιδεολογικά χέρια η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος, να υπενθυμίσω στην Επιτροπή μας ότι υπάρχει Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, που ασχολείται ε, από ε, την οπτική της γωνία με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακριβώς. Αναφέρομαι εδώ στο βραβείο Ζαχάροφ που ανέφερε ο συνάδελφος Ρινάλντι. Κύριε Πρέσβη. Όλοι θα ξέρετε ότι τα 30 χρόνια που συνεχίζεται αυτό το άνοιγμα της ε, Κίνας δίδεται μεγάλη σημασία στην ε, οικονομική πρόοδο, την ε, κοινωνική πρόοδο και στον εκδημοκρατισμό της Κίνας. Νομίζω ότι τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ε, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές και η μεγαλύτερη εξ όλων είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε στην κοινό, ο τρόπος σκέψης. Στο επίπεδο κράτος δικαίου, στο επίπεδο δημοκρατίας, σε επίπεδο προστασίας ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι όσοι από εσά είναι αντικειμενικοί μπορείτε να δείτε ε, πόση πρόοδος έχει γίνει στην Κίνα. Ε, στην περίπτωση του Χούτζα, ε, ο ίδιος ε, παραδέχτηκε ότι παραβίασε τον νόμο και τον αντιμετωπίζουμε με ανοιχτό, διαφανή, δημοκρατικό τρόπο. Επίσης, ε, δεν θα ξεχνάτε, τον τελευταίο χρόνο ε, στη σχέση μας με την Ταϊβάν έχει ε, σημειωθεί σημαντική βελτίωση. Αυτό βοηθάει όχι μόνο τους κατοίκους πέρα από τα... στην Ίσο, στην Ταϊβάν, πέρα από τα στενά δηλαδή, αλλά και σε μας. Ελπίζουμε επίσης ότι οι αρχές της Ταϊβάν θα αντιμετωπίσουν ε, με μεγάλη προσοχή την επίσκεψη του Δαλάη Λάμα. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι στις 5 Ιουλίου διοργανώθηκαν ε, κάποιες ε, εκδηλώσεις βίαιες εκδηλώσεις. Ελπίζουμε όμως ότι το ευρωπαϊκό κοινό θα αντιμετωπίσει τα γεγονότα της 5ης Ιουλίου με αντικειμενικότητα. Εμείς είμαστε κατά της τρομοκρατίας, κατά των αποσχιστικών τάσεων, αλλά βεβαίως θα σταματήσω σε αυτά τα σχόλια γιατί αυτά δεν έχουν σχέση με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Επανέρχομαι στα θέματα εμπορίου και οικονομίας. Καταρχάς, το εμπορικό έλλειμμα. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά ε, εξαγωγών για προϊόντα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα που εξάγεται προς την Κίνα από το 2004 μέχρι σήμερα αυξήθηκαν κατά 65%. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί λόγοι για την ε, έλλειψη ισορροπίας στο, ισοζύγιο πληρωμό, στο εμπορικό ισοζύγιο, αλλά κυρίως ε, η επανεγκατάσταση διαφόρων επιχειρήσεων, επενδυτικών και άλλων. Οι επιχειρήσεις που είναι κατεστημένες στην Κίνα κατασκευάζουν τα προϊόντα και τα πουλούν στην Κίνα. Και επομένως άλλαξαν τελείως οι ευρωπαϊκές εξαγωγές. Το 2006 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Κίνα Ε, έφτασαν σε επίπεδο εξαγωγών 206,6 δισεκατομμύρια ε, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τις κινέζικες εξαγωγές το 2006 ήταν 91,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο γύρο της Ντόχα το βασικό θέμα είναι η πολιτική βούληση να περάσει στις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό, να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις μέσα στα πλαίσια της εντολής που έχει ληφθεί και μέσα στο σημερινό πλαίσιο, ούτως ώστε να παγιωθούν τα αποτελέσματα και να επιληθούν τα υπόλοιπα εκρεμή θέματα. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα του γύρου της ε, Ντόχα θα πρέπει να λάβαν υπόψη τις ανησυχίες των αναπτυσσομένων κρατών θα πρέπει να υπάρχει προτιμησιακή και ειδική μεταχείριση και οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να δείξουν ευελιξία και να κάνουν περαιτέρω, να αναλάβουν περαιτέρω δεσμεύσεις για περαιτέρω μειώσεις. Επίσης για, την, για το αντι-dumping. Μέσα σε μια μικρή χρονική περίοδο υπάρχει μείωση των περιπτώσεων σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν συμπεριφέρονται σωστά, πραγματικά ε, εξετάζουμε αυτά τα θέματα, ε, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες παρά προβλήματα. Περισσότερο συνεργασία παρά ανταγωνισμός. Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προωθήσουμε τη συνεργασία, να αφήσουμε ανοιχτά κανάλια για επενδύσεις και για εμπόριο, να δημιουργήσουμε περισσότερες ε, ευκαιρίες επιχειρηματικές και πιστεύω ότι παρά την κρίση θα προχωρήσουμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα αντι-dumping. Επίσης, πιστεύω ότι θα ενδυναμώσουμε το διάλογο και χάρη στο διάλογο θα μειωθούν οι περιπτώσεις αντι-dumping. Χάρη στο διάλογο και φυσικά τη συνεργασία. Θέσατε και μία ερώτηση για τις ΕΠΑ, για τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης η Κομισιόν για αυτέ τι συμφωνίε και τι διαπραγματεύσει που γίνονται για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρική σχέση, όπω είπα και στη δική μου παρέμβαση, είμαστε λίγο απογοητευμένοι από πλευρά Κομισιόν, γιατί δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε όσο γρήγορα θα επιθυμούσαμε. Έχουμε τρία άρθρα, τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Τρία έχουμε συμφωνήσει από τα, τρία, από, από τα 20. Μετά από 1,5 χρόνο τα πράγματα δεν προχωρούν γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, προχωρούμε με τους Κινέζους. Υπάρχει δέσμευση από τους Κινέζους ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο και πιο γρήγορα το φθινόπωρο και ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε διάφορα άρθρα πριν φτάσουμε στη Σύνοδο Κορυφής του 2009. Κύριος Καζάκ, σας παρακαλώ οι βουλευτές να περιορίσουν ε, την εκφορά των ε, ερωτήσεών τους σε δύο λεπτά. Τόσο χρόνο έχουμε και στην Ολομέλεια. Σας παρακαλώ για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομο θα είμαι. Κύριε Πρέσβη, με μεγάλη χαρά άκουσα την παρέμβασή σας για τις διμερείς σχέσεις και πολυμερείς σχέσεις της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο και της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η διαπίστωση ότι και εσείς πλήδεστε από μέτρα και από πλευράς μας, αυτό δεν είναι σωστό. Μόνο 1% όλων των προϊόντων που εισάγονται πλήττονται από αυτά τα ευρωπαϊκά μέτρα. Και η έλλειψη ισορροπίας ε, στο εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ευρώπης και Κίνας ε, είναι δυσμενής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, πολύ σημαντικές για μένα. Πρώτον, τα μέτρα που την παραχάραξη και πειρατεία και πώς υπερασπίζεστε τα πνευματικά δικαιώματα. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος περιμένετε να σημειωθούν και άλλα βήματα προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης των προβλημάτων αυτών. Επίσης, τι δεσμεύσει θα αναλάβει η Κίνα ε, στην Σύνοδο κορυφή της Κοπενχάγης, ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δύο λεφτά ακριβώς. Έχετε μεγάλη εμπειρία με την τήρηση του χρόνου ο Κινέζος πρέσβης. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασία τους. Αυτό ακριβώς χρειάζεται η Κίνα για να μπορέσει να προωθήσει το δυναμικό καινοτομία της. Έχουμε ήδη ένα νομικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμμορφο με τους διεθνείς κανόνες. Επίσης, επιταχύνουμε τις προσπάθειες για να εφαρμόσουμε το νόμο. Ε, προβλέπουμε μάλιστα και ποινικέ ρήτρε στο νόμο. Και τον έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες εφαρμογής του νόμου. Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία μάλιστα να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό δείχνει το πόσο αποφασιστικοί είμαστε. Υπάρχει μια απόφαση ενός δικαστηρίου. Μία απόφαση που δείχνει την αποφασιστικότητα της Κίνας για να προστατεύσει τα δικαιώματα των δικαιούχων. Δικαιώματα ε, για την εκρίζωση ενός παρασίτου για ντομάτες κυπευτικές και, και άλλα κυπευτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο προσέλκυσε μεγάλη προσοχή από το διεθνή τύπο. Το θέμα γενικά των δικαιωμάτων νοματικής ιδιοκτησίας συζητείται πολύ συχνά. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί για αυτό το θέμα. Επίσης για την προστασία του κλίματος μας απασχολεί πάρα πολύ. Προσπαθούμε στα πλαίσια της κρατικής πολιτικής να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να επιτύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι η εθνική μας πολιτική. Και έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα για να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα καταρχήν και να επιτύχουμε τη μείωση των εργοβόρων επιχειρήσεων κατά 20%, δηλαδή να φτάσουμε στο 2010 στα νούμερα του 2005. Αν αυτό υλοποιηθεί, θα έχουμε μία μείωση των εκπομπών κατά ένα 1,5 ε, δισεκατομμύριο τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα είναι η πιο σημαντική συνεισφορά Παγκοσμίως, Επίσης, να κάνουμε διαθρωτικές ε, αλλαγές σε ενεργειακό επίπεδο. Στο οικονομικό μας πακέτο, πάνω από 300 δισεκατομμύρια γιουάν ε, σε επενδύσεις πηγαίνουν για την βελτίωση επιχειρήσεων ε, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Αν λάβουμε υπόψη μας τις ιστορικές ευθύνες που έχουν οι ανεπτυγμένες χώρες για μείωση των εκπομπών κατά 40% μέχρι το 2020 με βάση τα επίπεδα του 1990, νομίζω ότι εμείς έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε. Uh, Monsieur Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε από, τον, από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι υπήρχε ένας στόχος ε, για μια φιλόδοξη συμφωνία, λέει ο κ. Ζαντό. Δεν πρόκειται για ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, αλλά για διαπραγματεύσεις, για επενδύσεις και για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ερώτημα είναι προς την Κομισιόν. Μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και πότε για τη διαπραγμάτευση που έχει ήδη ξεκινήσει, για τα πεδία που έχουν καλυφθεί και για τους στόχους, τους εντός αγωγικών φιλόδοξους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμπροκειμένου. Τώρα και μια ερώτηση προς την ε, κινέζικη πλευρά. Στην ε, τελευταία παράγραφο του εγγράφου σας που μιλάτε για την πράσινη οικονομία και την ε, προστασία του κλίματος αναφέρεται κάποια ερωτηματικά ή κάποιες ανησυχίες ό,τι αφορά την τεχνολογική συνεργασία και τους περιορισμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σχετίζεται και με την Κοπενχάγη. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι, ευρωπαϊκές, οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί τους οποίους υπενήσεστε και ποιες είναι οι τεχνολογίες που εννοείται. Ε, πάντα στα πλαίσια της Κοπενχάγης. Η Κομισιόν θα σχολιάσει πρώτη. Ευχαριστώ. Όντως, είμαστε εν μέσω της διαδικασίας ε, για την σύνταξη του σχεδίου του κειμένου των διαπραγματεύσεων. Είναι σαφές που έγκυται το μείζον ενδιαφέρον στις βασικές επενδύσεις που αφορούν τις υπηρεσίες ε, και τις δημόσιες προημήθειες και τα TBTs, τα Technical Barriers to Trade, τεχνικά ε, εμπόδια στο εμπόριο. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που συζητούμε με την κινέζικη πλευρά. Όλα τα θέματα βρίσκονται επιτάπητος ε, στα πλαίσια των διαμαρτυρώσεων. Ορισμένα είναι πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά την επίτευξη πρόοδου από άλλα, αλλά φαίνεται σαφώς ποιο κομμάτι του κειμένου έχει συμφωνηθεί και ποιο όχι. Όπου περιμένουμε δηλαδή αντιπρόταση από την κινέζικη πλευρά. Και θα καταφτάσουν την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα. Κύριε Πρεσβευτά, ευχαριστώ. Η ό,τι αφορά τη συνεργασία για την υψηλή τεχνολογία, η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ε, τεχνολογία ε, στην ε, Κίνα. Και οποιαδήποτε θετική δεξιολήση στον τομέα βεβαίω είναι καλοδεχούμενη διότι ενδυναμώνει την ήδη έντονη συνεργασία μας στον τομέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτό που έλεγε ο κύριος Καζάκ και εγώ κάποια σχόλια, πρώτα απ' όλα υπόψη του περισβευτού, εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η κινέζικη πλευρά εργάζεται επί του θέματος της πνευματικής ιδιοκτησίας μας χαροποιεί διότι μέχρι τώρα είχαμε πρόβλημα πρόσβασης στην κινέζικη αγορά λόγω αυτού. Και θέλουμε να αρθούν τα εμπόδια που οφείλονται στην πνευματική ιδιοκτησία, στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σας υποστηρίζουμε και σας ευχόμεθα καλή επιτυχία σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας αυτή. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Εκτιμώ τις προσπάθειες που έχετε αναλάβει τα τελευταία χρόνια για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Το θέμα βεβαίω είναι ευαίσθητο και είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθείτε και με τον νάμα, ιδιαίτερα για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Έχετε στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία για τον άμα, γιατί η κοινή γνώμη στην Ολλανδία τουλάχιστον ενδιαφέρεται έντονα για το θέμα αυτό. Ο πρέσβης. Κοιτάξτε, ανέφερα και προηγουμένως τη θέση της κινέζικης κυβέρνησης ε, περί προστατευτισμού. Δεν θα υπέρ ουδήποτε μέτρο προστατευτισμού. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο θα ενισχυθεί περαιτέρω και βεβαίως θα γίνουν και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού. Μην ξεχνάτε όμως ότι όταν λέμε κοινό στην Κίνα μιλάμε για τρία δις ανθρώπους. Πάντως αυτή είναι η θέση μας, ε, την οποία επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει προστατευτισμός στη χώρα μου. Well, thank you. Φαντάστηκα ότι θα αναφέρεστε ε, σε θέματα φαρμάκων ε, στην Κίνα. Δεν έχω ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Θα το εξετάσω. Θα ε, εξετάσω τι νούμερα έχουμε. Αλλά στην φαρμακευτική βιομηχανία Έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά με την κινέζικη πλευρά. όσον αφορά την πρόσβαση νέων φαρμάκων στην ε, κινέζικη αγορά. Ε, ορισμένα συστατικά στοιχεία ορισμένων φαρμάκων κλπ. Υπάρχουν όμως όπως είπα στοιχεία τα οποία πρέπει να ψάξω πρώτα. Εσείς κύριε Μάρτιν. Επανέρχομαι στην ερώτηση που έγινε πριν για τους περιορισμούς σχετικά με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Μία από τις ανησυχίες της Ένωσης έχει και σχέση με την έλλειψη εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά την τήρηση των ε, συμφωνιών των ε, ε, δικαιωμάτων μηχανικής ιδιοκτησίας. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε στην εξαγωγή τεχνολογίας, κυρίως για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, εάν ε, γνωρίζαμε ότι θα τηρηθούν τα συμφωνημένα ή τέλο πάντων ε, οι ε, διεθνεί συνθήκε για την βιομηχανική διοκτησία. Επίσης, το θέμα της διακύμανσης του κινέζικου νομίσματος απέναντι στο αμερικανικό δολάριο αλλά και σε άλλα νομίσματα. Θα υποτιμηθεί το κοινωνικό νόμισμα. Καταλαβαίνω τους φόβους της Κίνας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πληθωρισμό. Αλλά πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ε, ελλείψης ισορροπίας στο ισοζύγιο και γενικότερα να ενθαρρυνθεί, ε, να, ενισχυθεί η, οικονομική, η διεθνής οικονομική ανάπτυξη. Και για το Hong. Kong. Έχουν γίνει αλλαγέ και στο Χογκόνγκ και στην Κίνα. Κινείστε προ την κατεύθυνση ενό ενιαίου οικονομικού συστήματο στην Κίνα και στο Χογκόνγκ ή θα επιτρέψετε την ύπαρξη δύο διαφορετικών συστημάτων. Ο πρέσβης. Όπως είπα, η προστασία ε, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδίω για, το, το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ελπίζω ότι θα είναι το επόμενο βήμα. Και οι δύο πλευρές θα κάνουν βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι σημαντικός τομέας. Δεύτερο, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Από τον Ιούλιο του 2005, όταν Ε, η στο 21,1%, 1,8% και 0,3% απέναντι στο αμερικανικό δολάριο, στο ευρώ και στο ιαπωνέζικο γεν. Άρα πρόκειται για μια διακύμανση ε, προς δύο κατευθύνσεις. Εμείς ε, το μετρούμε πάντοτε απέναντι σε ένα καλάθι νομισμάτων για τη διακύμανση του νομισματός μας και σε ό,τι αφορά την ε, ζήτηση και προσφορά στην αγορά. Έχει ενισχυθεί η ζήτηση του νομίσματός μας και αυτό έχει ενισχύσει την διακύμανση. Η κινέζικη κυβέρνηση όμως θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις αλλαγές στις δοκιμάνσεις ε, βασικών ε, διεθνών νομισμάτων για να διατηρηθεί μια βασικά σταθερή ε, συναλλαγματική ισοτιμία. Τώρα για το Χονγκ Κόνγκ. Από το 1997 έχουμε μία χώρα και δύο ε, οικονομικά συστήματα. Αυτή είναι η πολιτική, όχι μόνο βέβαια στον πολιτικό τομέα, αλλά και ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα και αλλού, στο Χονγκ Κονγκ, ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα του Χονγκ Κονγκ. Είτε και στην ε, οικονομική κρίση τότε του 1997, αλλά και σε τούτην εδώ που ζούμε τώρα. η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας και στις δύο αυτές περιπτώσεις έπραξε πάντο δυνατό για να διατηρήσει την ε, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ είναι σταθερό, η οικονομία του βελτιώνεται. Αυτά θέλω να σας πω. Μα είναι και το Μακάο που ήταν πορτογαλικό. Ο κύριος Σαρίφ. Euh, Ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τα όσα είπε ο Κινέζος πρέσβης, καθώς και αυτά που είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Αυτό που είναι ενδιαφέρον ε, όταν μιλάμε για εμπόριο είναι το κοινωνικό dumping και ο σεβασμός των ε, κοινωνικών κανόνων. Η, ο μη σεβασμός συνδέει και αυτή η ανισορροπία που ανέφεραν οι συναδελφοί μου παίζουν ένα μεγάλο ρόλο γιατί το αντι-dumping οδηγεί στο μη σεβασμό διαφόρων κανόνων. Θα ήθελα να μου πει ο πρέσβης τη γνώμη του για το θέμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την συνδικαλιστική ελευθερία στην Κίνα, για την αναγκαστική εργασία, για την παιδική εργασία για την αξιοπρεπή εργασία, για τον ε, σεβασμό των κανόνων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, σημαντικότατα θέματα και για τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Παρά το γεγονός ότι υπογράφηκε μια συμφωνία τον Ιανουάριο για το θέμα της εργασίας, παρά την ε, συμφωνία αυτή που υπογράφηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, ε, μοιάζει να μην έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στο θέμα της εργασίας ε, το τελευταίο διάστημα. Τι σκοπεύει να κάνει η κινέζικη κυβέρνηση για όλα αυτά τα θέματα, για τους κοινωνικούς κανόνες, υπό την ευρία έννοια του όρου. Thank ξέρετε, η Κίνα έχει πληθυσμό 1,3 δις έχει πολλές ανισότητες, είμαστε ακόμα στα ημίσια του δρόμου που οδηγεί στην εκβιομηχάνηση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω του όγκου του πληθυσμού μας είναι βεβαίως σημαντικά. Η κινέζικη κυβέρνηση πάντως προσπαθεί να εφαρμόσει αυστηρά μέτρα και νομίζω ότι έχουμε επιτύχει κάποιους από τους στόχους της ε, χιλιετίας εις ό,τι αφορά τη μείωση της στόχιας που μειώθηκε από 200 εκατομμύρια, από 250 εκατομμύρια σε 11 εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα πολλοί πολίτες που ζουν με ένα ή λιγότερο δολάριο την ημέρα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και το θέμα αυτό, πράγμα το οποίο προσπαθούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα λάβετε υπόψη σας αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα τα πληθυσμιακά ε, δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε λέει η κυρία Σαρνές. Κύριε Πρέσβη, δεν είμαστε ίσοι στο ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο, γιατί δεν σεβόμαστε τους ίδιους κανόνες. Είτε υγειονομικούς, είτε περιβαλλοντικούς, είτε εμπορικούς. Και αυτό μας προσάπτουν οι πολίτες μας με το λεγόμενο κοινωνικό και περιβαλλοντικό dumping. Θα ήθελα λοιπόν την ειλικρινή σας ή δυνατόν για το πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα. Η πρώτη προσέγγιση είναι να βάζουμε φράγματα για να προστατευόμαστε. Εμείς έναντι άλλων που έχουν κοινωνικό dumping. Και ο δεύτερος τρόπος είναι εσείς να προσπαθήσετε να συγκλίνετε ή να προσεγγίσετε τα δικά μας πρότυπα. Θα ήθελα την ειλικρινή σας άποψη από αυτό. Και κάτι ακόμα. Δύο τινά. Πρώτο, εις ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας ε, των ε, μισθωτών, των εργαζομένων στην Κίνα και τα παιδιά, θα επικυρώσετε τις διεθνείς ε, συμβάσεις, τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Και δεύτερο, για την Κοπενχάγη, είπατε όντω στα προκαταρκτικά σα σχόλια ότι δεν μπορείτε να καταπολεμήσετε πλήρως τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπλοκάρει κάποιες, ε, κάποια μέτρα ε, μεταφοράς τεχνολογίας. Και κάποιο άλλο συνάδελφο ρώτησε και επαναλαμβάνω και εγώ. Πού ακριβώ αναφέρεστε. Κυρία Σαρνές λέει ο πρόεδρος, θα ήθελα να απαντήσει τώρα ο πρέσβης και μετά να σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα του αθέμη του ανταγωνισμού, διότι περί αυτού πρόκειται, αν κατάλαβα καλά, ο πρέσβης. Ευχαριστώ. Η κινέζικη κυβέρνηση, όπως είπα, έχει θέσει σε ισχύ ένα νομικό πλαίσιο για τις συνθήκες εργασίας και την εργασία των παιδιών, των ανηλίκων παιδιών. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, είναι όμως σποραδικά και αφορούν από μεμακρυσμένες και δύσκολα ελέγξιμες περιοχές. Τώρα, για τον αθέμητο λεγόμενο ανταγωνισμό, δηλαδή το ότι δεν ξεκινάμε από την ίδια βάση. Ίσως να μην γνωρίζετε ότι πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε είναι υψηλής ποιότητος και ε, χαμηλής ε, τιμής που παρασκευάζονται στην Κίνα. Μην κοιτάζετε λοιπόν το θέμα μονομερός δεν είναι μόνο εμπορικό. Υπάρχουν και άλλες πτυχές. Η Κομισιόν η ε, βιώσιμη ανάπτυξη και οι συνθήκες εργασίας είναι άρρηκτο κομμάτι των ε, διαπραγματεύσεων. και αφορά τι διαπραγματεύσει των συναδελφών μα από, τις, ε, από Εξωτερικών Σχέσεων και την ε, κινέζικη πλευρά. Από πλευράς ε, εμπορίου για τις ΕΠΑ κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου πάντα και στα πλαίσια αυτά εξετάζουμε τα πορίσματα της μελέτης αυτής σε μεγάλο βάθος. Η σχετική μελέτη έχει συνταχθεί από ε, εξωτερικό σύμβουλο και είναι διαθέσιμη ε, και πρόσβασιμη σε όλους. Τελευταίο ερώτημα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ερώτημά μου απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Κίνα είναι ο βασικότερος εμπορικός μας εταίρος. Και είπε ότι η μέση τάξη αυξάνεται και πληθύνεται και ίσως γιατί μπορεί να αγοράσει περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ερώτημα προς την Κομισιόν. Πώς συμφιλιώνεται την όθηση που δίνεται στην Κίνα να φτάσει σε επίπεδα οικονομίας της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα διακρίνεται μέτρα πρωτοτευτισμού και παρεμβατισμού του κράτους. Η ιδιωτικοποίηση που τόσο επίμονα ενθαρρύνεται είναι, έχει τραγικά αποτελέσματα για την ευημερία των πολιτών και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σε ένα χαλιβουργείο το, με, το Μάιο χάθηκαν 20.000 θέσεις εργασίας σε σύνολο 35.000. Ε, θα χανόντουσαν μάλλον ε, εάν δεν αναλάβαναν συνδικαλιστική δράση ε, οι εργαζόμενοι. Τέτοια φαινόμενα απαντώνται ε, πάρα πολύ συχνά και αυτά απορρέουν από τα μέτρα ιδιωτικοποίησης αυτών των επιχειρήσεων. Κομισιόν, λοιπόν, όταν ακόμα, ακόμα όταν πριτανεύουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, όταν θέλετε να προστατεύσετε ε, τις ευρωπαϊκές ε, ε, ε Πώς είναι δυνατόν να μιλάτε συγχρόνως για περισσότερη ιδιωτικοποίηση, για οικονομία της αγοράς, όταν τα αποτελέσματα είναι τραγικά για τις συνθήκες εργασίας του Κινέζου εργαζόμενου, που είναι από τις χειρότερες στον κόσμο. Το γκούλαγκ του σταλινισμού. Αυτό το πρόσωπο έχει σήμερα στην Κίνα. Τι γίνεται με τα συνδικάτα. Τι γίνεται με την προστασία των εργαζομένων. Έναντι της προστασίας τους από αυτό το χήμαρο εξελίξεων που είναι αρνητικό ενώ που είναι η παγκοσμιοποίηση. Uh, Για το καθεστώς ε, οικονομίας της αγοράς. Δεν νομίζω ότι η Κομισιόν πιέζει την Κίνα να αποκτήσει αυτό το καθεστώς. Νομίζω ότι η κινέζικη κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση και επιθυμεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο οικονομίας της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποίησεις, και αυτό είναι πολιτική της κινέζικης κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ή μπορεί η Κομισιόν να πιέσει ε, την Κίνα και να της επιβάλλει κάτι τέτοιο. Καλύτερα θα ήταν να απαντήσει όμως και ο Κινέζος πρέσβης ε, σε αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες ε, που λειτουργούν στην Κίνα, πολλές από αυτές είναι πολύ δραστήριες σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά και εργατικά πρότυπα και πολλές από αυτές έχουν καλά πρότυπα στο εσωτερικό τους και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να λέμε ότι επειδή είναι επιχειρήσεις από οικονομίες της αγοράς, για αυτό το λόγο αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ε, ε, χειρότερα από ό,τι θα τις αντιμετώπιζαν οι κρατικές ε, εταιρείες. Φυσικά υποστηρίζουμε τη συζήτηση για την κοινωνική ευθύνη με τις εταιρείες μας στην Κίνα. κάναμε και πολλά σεμινάρια για αυτά τα θέματα. Η συζήτηση συνεχίζεται. και στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, αλλά και στους, στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, στη Ρελέξ δηλαδή, μαζί με την κινέζικη κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Helen Koenig που ήρθε εδώ από πλευράς Κομισιόν και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Κινέζο πρέσβη που ήρθε σήμερα στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Όπως είπα και στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε τις σχέσεις με την Κίνα εμείς ως ε, ομάδα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα στείλουμε εκπροσώπους στη Γενέβη για την Υπουργική Σύνοδο. Νομίζω τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα γίνει. Θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε τότε να συναντηθούμε με τον Υπουργό Εμπορίου στη Γενέβη ή να διευκολύνεται μια τέτοια συνάντηση, κύριε Πρέσβη, με τον Υπουργό. Και το τελευταίο. Ίσως είναι υπερβολικό το αίτημα, αλλά η Επιτροπή μας εξετάζει το ενδεχόμενο αιτήσεων επισκέψεων ε, σε διάφορες χώρες. Ίσως στο μέλλον θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε την Κίνα. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά που ήρθατε. Και σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Πολύ ωραία. Πάμε στο σημείο 12. επιπτώσεις της ε, <clears throat> οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στο διεθνές εμπόριο. Ας περιμένω λίγο να αδειάσει η αίθουσα και εν συνεχεία να μιλήσει ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν για το σημείο αυτό. Impact of economic and financial crisis situation on international trade. I think it's... Λοιπόν, σημείο 12. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση. Ακούσαμε τον Κινέζο πρέσβη να περιγράφει την κατάσταση ε, και πώς επηρεάζεται και η Κίνα. Ε, η κρίση αυτή, η οικονομική και χρηματοπιστωτική, είναι πολύ έντονη και στην Ευρώπη και στη δική μου χώρα ειδικά. Νομίζω ότι είναι ένα επίκαιρο θέμα που απευθύνομαι προς την Κομισιόν ε, να μας πει πώς βλέπει το μέλλον. Ε, πάντα πίστευα ότι αν ρυθμίσουμε την τόχα θα βοηθήσουμε για να εξέλθουμε από την κρίση. Αλλά νομίζω ότι όλες οι εμπορικές σχέσεις με οποιαδήποτε χώρα θα βοηθούσαν θα βοηθούσε για να αυξηθούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω τα προβλήματα απασχόλησης. Μειώνται η θέση απασχόλησης όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να μας διαφωτίσει η Κομισιόν για ό,τι συμβαίνει. Να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε και σας και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ για την εκλογή σας ή επανεκλογή σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτή την ε, κοινοβουλευτική θητεία, καλή επιτυχία σε εργασίες της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Και εκ μέρους της Κομισιόν σας ε, διαβεβαιώ ότι θα σας υποστηρίξω σε εργασίες σας. Να πω δύο λόγια για μένα. Είναι η πρώτη μέρα ως βασικός, ε, πρώτη μου μέρα ως βασικού οικονομολόγου στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και μου έλαχε να έρθω εδώ και να μιλήσω για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας. Πολύ σύντομα να πω δύο λόγια για τη μονάδα βασικών οικονομολόγων στην ε, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ο βασικός μας ρόλος είναι να κάνουμε μια υψηλού επίπεδου οικονομική ανάλυση ε, για τις διάφορες εμπορικές πολιτικές που έχουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη Γενική Διεύθυνση για να αξιολογήσει την επίπτωση των πολιτικών ανά τον κόσμο και να θέσει προτεραιότητες για νέα μέτρα εμπορικής πολιτικής. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με συναδέλφους από άλλες μονάδες και προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές πτυχές διαφόρων μέτρων εμπορικών πολιτικών. Επίσης, είμαστε σε επαφή με άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν για να απλουστεύσουμε άλλους τομείς. Παραδείγματος χάρη στην τομέα της παγκοσμιοποίησης ή του ανταγωνισμού προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι από πλευράς εμπορίου, από τη σκοπιά του εμπορίου, το εμπόριο παίζει το ρόλο του και σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια διαφάνεια. Ε, εξετάζουμε τις τελευταίες στατιστικές και τις δίνουμε και στους συναδέλφους και στα άλλα όργανα, αλλά και στο κοινό και στην κοινωνία των πολιτών. Ε, είμαστε εστιακό σημείο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Ε, παρακολουθούμε και παρακολουθήσαμε από την αρχή τις επιπτώσεις ε, της κρίσης ε, στο εμπόριο και στις εμπορικές πολιτικές και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής για να απαντήσουμε ε, σε αυτές τις προκλήσεις και να βγούμε από την κρίση. Λοιπόν, για να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, θα ήθελα να σας περάσω καταρχάς τρία βασικά μηνύματα. Θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, βασικές εμπορικές παραμέτρους της κρίσης. Εν συνεχεία θα μιλήσω για τις πολιτικές που έχουμε προωθήσει μέχρι τούδε και κάποιες σκέψεις για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Για να περιγράψω την κρίση θα την περιγράψω με τρεις λέξεις. Ήταν ξαφνική, α, σοβαρή και συγχρονισμένη. Ευνίδια γιατί τους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου ε, σε τήσια βάση ε, έπεσαν οι εξαγωγές κατά 40%. Ε, ήταν δραματικό γιατί οι περισσότεροι ε, εκτιμητές δεν το περίμεναν. Ε, γιατί ε, από πολλές πλευρές ήταν μεγαλύτερη και από το κράκτη 29. Θα σας το αποδείξω αυτό το σημείο. Και επίσης από τον Νοέμβριο του 2008 Είχαμε μία μείωση κατά 342 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στα, στο εμπόριο των ε, εμπορευμάτων. Αυτό θα σήμαινε ότι η Γαλλία, η, Ιταλία είχε χάσει όλες τις εξαγωγές της μέσα στο 2008. Ε, η Πολωνία, ας πούμε, σαν να έχει χάσει όλες τις, ε, όλα τα κέρδη από τις εξαγωγές. Αυτό είναι έτσι μια μια παραβολή για να σας βοηθήσω να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Κάτι πολύ σημαντικό για την κρίση είναι ο σύγχρονος χαρακτήρας της κρίσης. Δηλαδή σχεδόν όλες οι χώρες την ίδια χρονική στιγμή επλήγησαν την κρίση. Ε, κανένας δεν δραπέτευσε για πρώτη φορά Καμία ε, αγορά δεν παρέμεινε ακέραιη ως ε, τελευταία καταφυγή για εξαγωγές. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό φαινόμενο. Ε, διαφορετικό από αυτό που συνέβη σε άλλες κρίσεις με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα σας αναφέρω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Μπορούμε να επανέλθουμε αν έχετε ερωτήσεις. Με αυτή τη γραφική παράσταση θέλω να πω κάποια πράγματα. Πρώτον, ο κόσμος το 2009 ε, θα βρίσκεται σε ύφεση, θα υπάρχει αρνητική ανάπτυξη συνολικά. Ε, μείον 1,5% είναι η πρόβλεψη, που είναι αρκετά σημαντικό. Ε, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα βγούμε από την κρίση. Αν το, πρέπει να το λάβουμε υπόψη να δούμε πώς θα βρούμε, βγούμε από την κρίση. Επίσης, η κρίση δεν έπληξε όλες τις οικονομίες με τον ίδιο τρόπο. Κυρίως έπληξε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, Ιαπωνία, τη ΣΥΠΑ, τις αναπτυγμένες δηλαδή οικονομίες πολλές αναπτυσσόμενες ε, και αναβιώμενες οικονομίες, ειδικά και η Κίνα, παρότι επλήγησαν από την κρίση, θα έχουν θετικές αναπτύξεις ε, το 2009. Και το 2010 η ανάπτυξή τους ήταν αρκετά μεγάλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παγκόσμιο εμπόριο είναι σε καλή κατάσταση. Το 2009 ο ΠΟΕ προέβλεψε μείον 12% και του χρόνου θα υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη κατά 1% στο παγκόσμιο εμπόριο. Για την Ευρώπη, η γραφική παράσταση δείχνει ποια ήταν τα επίπεδα του 2005. Η κρίση μας έφερε πίσω σε αυτά τα επίπεδα. Όλη η ανάπτυξη που υπήρξε από το 2005 μέχρι τούδε εξαφανίστηκε, ξανεμίστηκε και φτάνουμε πάλι στα επίπεδα του 2005, σαν να μην είχαμε κουνηθεί καθόλου από εκεί. Ε, το 2000, το 2009 που βρίσκεται στην κόκκινη γραμμή, ε, βρίσκεται πολύ πάνω στην αρχή από τα επίπεδα του 2005 αλλά περίπου στα επίπεδα του 2005 στη συνέχεια του έτους. Υπάρχει μια κάμψη. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ταυτόχρονη εμφάνιση της κρίσης σημαίνει ότι οι εξαγωγές στις βασικές ε, οικονομίες ακολουθούν παράλληλες ροές. Ε, από τον Νοέμβριο οι εξαγωγές ε, μέχρι και κάνα δύο μήνες πριν είδα σε ελεύθερη πτώση. Υπάρχουν όμως ε, κάποια σημάδια αισιοδοξία. του τελευταίους δύο-τρεις μήνες ε, υπάρχουν κάποια σημάδια ανάκαμψης. Βλέπουμε τις πρώτες, ε, τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι τον πιάσαμε τον πάτο και τώρα έχουμε πάρει την ανιούσα σε επίπεδο εμπορίου. Για το θέμα της ανάκαμψης θα πρέπει να δούμε χωριστά τις τιμές και τους όγκους. Το βασικό που πρέπει να είμαστε σίγουροι είναι ότι αυξήθηκαν οι όγκοι. Οι τιμές σε καθημερινή βάση μπορούν να δικημένονται. Το βασικό είναι να ανακάμψουν οι όγκοι. Αυτό είναι ο βασικότερος δείκτης για το εμπόριο. Και με βάση τις στατιστικές, ε, το παγκόσμιο εμπόριο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ξανά. Θα υπάρξει ανάκαμψη, παρόλα αυτά δεν πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί. Εγώ εδώ σας δείχνω ποια ήταν η εξέλιξη της, στα πλαίσια της μεγάλης ύφεσης του 29 ε, για το εμπόριο. Ε, με το μπλε είναι η εξέλιξη σήμερα και με το ροζ η εξέλιξη τότε. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει διπλή πτώση. Η κυρία Μέρκελ ε, μίλησε χθε για στρατηγικέ που μπορεί να είναι πολύ απότομε και που μπορεί να θέσουν να αμφιβόλω την παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί από τη γραφική παράσταση του, 2000, 1929, ε, ότι μετά την ελεύθερη πτώση υπήρξαν κάποιοι μήνες ε, ανάκαμψης. Και ο κόσμος πίστεψε ότι βγήκε από το τούνελ, αλλά μετά από λίγο ξανά πέσε πάλι ε, η οικονομία. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Θα πρέπει να μάθουμε τα μαθήματα από το παρελθόν, να αποφύγουμε τα λάθη για να... και να εστιάσουμε στις εμπορικές πολιτικές ε, με στεναρό τρόπο. Το μήνυμα είναι πολύ απλό. Σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις πρέπει να δώσουμε με τις εμπορικές πολιτικές, το εμπόριο είναι τμήμα της λύσης, δεν είναι τμήμα της κρίσης, δεν είναι το εμπόριο που προκάλεσε, αυτό που προκάλεσε την κρίση, είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που μπορεί να επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη αντίθετα. Και το απλό μήνυμα ποιο είναι λοιπόν. Πράγματα τα οποία γνωρίζαμε στο παρελθόν. Και πάντα ήταν ε, τμήμα της ε, εμπορική μας πολιτικής εδώ και πολλές δεκαετίες. Πρέπει να αποφύγουμε τον προστατευτισμό. Οι χώρες δεν πρέπει να καταφύγουν εκεί. Ο προστατευτισμός θα μας οδηγήσει σε μια μεγάλη ύφεση. Η κρίση θα επιταχυνθεί, Υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων η Κομισιόν και άλλοι εταίροι ανά τον κόσμο ε, προσπαθούν να βοηθήσουν τα πράγματα. Ανοιχτές αγορές. Οι ανοιχτέ αγορές και ο μηχανισμός του ΠΟΕ ε, βοήθησε του πρώτους μήνες μετά την κρίση. Κατά τη διάρκεια τη μεγάλης ύφεση ε, δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός, δεν υπήρχε δυνατότητα να κρατηθούν οι δασμοί κάτω από ένα ορισμένο κατόφλι. Ε, τώρα έχουμε τέτοιου κανόνες ε, για τον προστατευτισμό, για, τις, ε, για τους δασμούς, για τις επιδοτήσεις, για τις δημόσιες προμήθειες. υπάρχουν όμως ακόμα κάποια παραθυράκια τα οποία πρέπει να καλύψουμε και το G20 πήρε κάποιες δεσμεύσεις για όλα αυτά τα θέματα. Το G20 προσπαθεί να προωθήσει το πακέτο κινήτρων ε, στα πλαίσια χωρών που βρίσκονται περίπου στην ίδια κατάσταση, εντυγμένων χωρών. Όλα αυτά τα μέτρα τα προωθήσαμε και με αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε το χειρότερο σενάριο στη σημερινή κρίση. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, είμαστε ε, το, ο πρώτος εμπορικός ε, όμιλος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ε, υπηρεσίες, τα αγαθά, αλλά και τις επενδύσεις. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη στο να κρατήσουμε αγορέ, τις αγορές μας ανοιχτές και μην ξεχνάμε ότι τα δύο τρίτα των εισαγωγών μας τελικά καταλήγουν ως εξαγωγές. Επομένως, να μην κρατάμε μόνο τις... Είναι σημαντικό να κρατάμε τις αγορές ανοιχτές, ε, και την εσωτερική αγορά αλλά και τις ε, εθνικές αγορές. Γιατί είναι πολύ εύκολο να διαταραχθούν από μέτρα προστατευτισμού αυτές οι αγορές που αποτελούν μια λυσίδα ούτως ή άλλως οι αγορές. Και η διατάραξη των, της λειτουργίας των αγορών είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ε, το διεθνές εμπόριο έχει παγκόσμια φύση. Αν διαταραχθούν οι εμπορικές ροές, επηρεάζεται το ΑΕΠ σε πάρα πολλές χώρες, ε, με ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας. Τώρα, συμπερασματικά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εν συνεχεία. Χάρη στους δύο μηχανισμούς που ανέφερα προηγουμένως. Και κάτι άλλο. Στο γεγονός ότι η Κομισιόν πρόθεσε κάποιους μονομερείς μηχανισμούς, την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι χώρες ανταποκρίθηκαν στην κρίση, ούτως ώστε οι απαντήσεις να μην είναι προβληματικές, να μην προωθούν τις διακρίσεις στο εμπόριο. Δηλαδή, με τον, με τους με τον πολυμερή μηχανισμό, με τον ΠΟΕ, ε, με το G20 και με τα μέτρα της ευρωπαϊκής πολιτικής, ε, έχει μειωθεί σημαντικά η τάση για προστατευτισμό και έτσι αποφύγαμε το χειρότερο σενάριο. Τους περασμένους μήνες είδαμε ότι το σύστημα του ΠΟΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε αναθεωρηθεί η Ντόχα στο Πίτσμπουργκ είτε όχι. το γεγονός ότι υπάρχουν ε, κάποια πρώτα στεναρά σημάδια ε, ανάκαμψης, αυτό δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να μειώσουμε τις προσπάθειες. Επίσης θα πρέπει να επανατονίσουμε τη σημασία μας ε, στον DDA, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μας βοηθούν για να προωθήσουμε την τόχα. Με μείωση του προστατευτισμού, των ε, δασμών κτλ. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, αν με επιτρέπετε, λέει ο Πρόεδρος. Μιλήσατε για τον τρόπο με τον οποίο τούτη εδώ η κρίση θυμίζει εκείνη την παλαιά της δεκαετίας του 2030. Εγώ θεωρώ ότι υπήρξε μια ε, βαθύτατη έλλειψη ευθύνης ορισμένων πιστοτικών ιδρυμάτων στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν ε, στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές με κυρίως τα δάνεια που χορηγήθηκαν για τις αγορές ε, κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος είναι υπεύθυνο εν τέλει για την σώρευση αυτών των χρεών. Γιατί νομίζω ότι τελικά δεν έχει εξηγηθεί αυτό. Εγώ θεώρησα ότι η Κομισιόν θα είχε κάποια σχέση, θα είχε ε, την ικανότητα να κατανοήσει με ποιο τρόπο λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και η γνώμη μου είναι, αν και ίσως κάνω λάθος, ότι όσοι ε, συμβούλευαν τις τράπεζες και τα άλλα ιδρύματα να αγοράζουν τα χρέη αυτά, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι συσσωρεύοντας τα χρέη αυτά ρίχνουν λάδι σε μια φωτιά η οποία τελικά θα καταβολθεί τα πάντα. Δεν θα έπρεπε η ε, Κομισιόν να είχε προτείνει κάποια ε, νομοθεσία. Εγώ βέβαια δεν είμαι υπέρ να φορτώνονται οι αγορές με ε, νομοθεσίες, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε συσταθεί στις τράπεζες να αποφύγουν να αγοράζουν τα χρέη αυτά. Δεν υπήρχε κάποια ευθύνη προκειμένου. Άσκησαν την απαραίτητη επιμέλεια. Εγώ νομίζω πως όχι. Ο εμπειρογνώμων. Μίλησα για trade, εμπόριο, εμπορική πολιτική δεν καλύπτω εδώ το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα της δραστηριότητες των λεγόμενων hedge funds ή άλλων διαμεσολαβητών. Αλλά έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπήρξαν παραλήψεις ε, στο ε, κανονιστικό σύστημα σε όλο τον κόσμο και σε άλλους σημαντικούς ε, εταίρους, όχι μόνο στην Ευρώπη και γνωρίζετε μάλλον καλύτερα και από μένα τις ε, δεσμεύσεις που ειχαν λαβει αναλάβει G20 και τις συνεχιζόμενες ε, συζητήσεις και τη σημασία που έχει το θέμα αυτό στην ατζέντα του G20. Εγώ δεν θέλω να κρίνω το αποτέλεσμα της διάσκεψης αυτής της κορυφής, αλλά σίγουρα ένας από αυτούς, ε, αυτά, αυτά που λέτε είναι ένας από τους λόγους που ξεκίνησαν την παγκόσμια οικονομική κρίση, που την οδήγησαν να, να την προκάλεσαν. Θα έπρεπε μια τέτοια κρίση όντως να είχε προβλεφθεί και να είχε μετριαστεί με αυστηρότερους ελέγχους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλή ερώτηση. Τι γίνεται όταν ε, α, μια αγορά στις ΗΠΑ Υπάρχουν ορισμένες, ε, υπήρχαν ορισμένες ενδείξεις ότι μπορούσε να γίνει το φθινόπωρο φέτος. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτησή σας. Δεν ήταν απόλυτα σαφής. Για ποια αγορά μιλείτε. Ε, από άψη όγκου η CDS Market είναι παρόμοια με την ε, αγορά υποθηκών, εν υποθηκών δανείων. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω πριν ότι όταν ξεφεύγουμε από το στενό φάσμα της εμπορικής πολιτικής ή εν πάση περιπτώσει των όσων ε, θεμάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένα, άλλα πράγματα θα έχουν κάποια ε, επιρροή στη, ε, στη μακροοικονομική σταθερότητα. Αλλά αυτό που ρωτάτε ξεφεύγει από, αν θέλετε, το χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων μου. Αλλά συμφωνώ μαζί σας και επαναλαμβάνω αυτό που απάντησα και στον πρόεδρο. Ε, υπάρχουν ορισμένε ψηφίδες που πρέπει να μπουν σε σωστή θέση για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες στο παγκόσμιο επίπεδο μπορούν, να είναι καλύτερα σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα όχι μόνο για τις επενδύσεις και το εμπόριο αλλά και για την ε, ε, χρηματοδότηση. David, εσείς. Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τώρα για το γράφημά σας που δείχνει την προσωρινή εκείνη ανάκαμψη ε, για τρεις-τέσσερις μήνες ε, στην ε, κρίση του 1930 και μια παρόμοια που φαίνεται τώρα. Αυξάνουν οι τιμές των πρώτων υλών, αυξάνουν οι τιμές των μεταποιημένων προϊόντων είτε οφείλεται η αύξηση των τιμών στο ότι μειώνονται τα αποθέματα πρώτων υλών και αρχίζουν και πιέζονται οι τιμές προς τα πάνω. Και σχετικό ερώτημα. Για μήνες μιλούμε για την παγκόσμια κρίση, τα τρόφιμα. Η παρούσα κρίση πώς επηρεάζει την αγορά τροφίμων σύμφωνα με τις στατιστικές σας. Υπάρχει μια κίνηση των επενδυτών από τη βιομηχανία προς την ε, ε, γεωργική οικονομία και προσπαθήστε λίγο να μαντέψετε. Είχαμε εδώ κοντά μας τον κύριο Σάλιβαν χθε που είπε ότι τα προστατευτικά ανακλαστικά δεν ήταν τόσο σημαντικά ανακλαστικά μέχρι τώρα όσο φοβούνταν ορισμένοι. Δεν έχουμε όμως ακόμα και στοιχεία για την, ε, ε, για την απασχόληση. Κατά πόσο επλήγει η απασχόληση δηλαδή. Τι στοιχεία έχετε εσείς και η ενδεχόμενη αύξηση της απασχόλησης, τι συνέπειες θα έχει στη, στα προστατευ... προστατευτισμό, δηλαδή στα αναγκαστικά προστατευτισμό. Σημαντικές ερωτήσεις. Μίλησα πριν για την ε, κίνηση των τιμών απέναντι στην κίνηση των όγκων. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα ότι βλέπουμε τα πρώτα ε, στοιχεία μιας ανάκαμψης. Δεν μίλησα βέβαια πριν για τις τιμές. Οι τιμές πιέζονται και από μια πίεση των τιμών ε, στις πρώτες ύλες που πέρασαν από ένα ιστορικό ε, χαμηλό μετά από ένα ιστορικό υψηλό που ε, ήταν πριν. Και επίσης πράγματι για την κρίση των τροφίμων δεν την ακούμε τώρα τόσο πολύ γιατί οι τιμές για τα αγαθά αυτά έχουν μειωθεί, όχι όλες, όμως δεν έχει μειωθεί η ζήτηση για ε, βασικά τρόφιμα και η ζήτηση είναι ένας παράγοντας που ε, εξηγεί τις, ε, τις βασικές επιρροές στη, στο εμπόριο. Δεν σταμάτησε ο κόσμος να χρειάζεται καθημερινά τρόφιμα οι τιμές των εξαγωγών έχουν ε, μειωθεί πολύ περισσότερο από την, ε, ε, τις εισαγωγές. Στην τρίτη σας ερώτηση, τα επίπεδα της ανεργίας θα αυξηθούν λίγο στους επόμενους μήνες. Έχουμε ήδη κάποια πρώτα στοιχεία για την ανεργία στην Ευρώπη, ήδη διψήφια ποσοστά. Η ανεργία θα διατηρηθεί περισσότερο από ό,τι θα μπορέσει να αποδώσει η, η θεμελιώδης ανάκαμψη. Πάλι όμως, μία ανάκαμψη που να βασίζεται σε εξαγωγές είναι σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για άλλες ε, χώρες οι οποίες εξαρτώνται από μεγάλες ε, αγορές προς τις οποίες γίνονται εξαγωγές. Και βεβαίως για να εξασφαλίζουν το εισόδημα που είναι απαραίτητο για, να, ε, για την αγορά των ε, ε, βασικών αγαθών. Και αν οι τιμές παραμείνουν στα παρόντα επίπεδα, βρίσκονται σε ένα επίπεδο όπου δεν επιτρέπει να μιλούμε για μια κρίση στην αγορά των τροφίμων. Είναι δηλαδή σε αρκετά καλό επίπεδο. Ήταν 200, 200 ευρώ ο τόνος τα δημητριακά πριν από 18 μήνες και σήμερα είναι στα 70 ευρώ ο τόνος. Αυτό το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον. Κύριε Ζαντώ, ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Αν συνοψίσω σχηματικά ε, την παρέμβασή σας λέτε το εμπόριο δεν είναι η αιτία της κρίσης αλλά τμήμα της ε, λύσεως Αυτή η θεώρηση των πραγμάτων σημαίνει ουσιαστικά ότι θεωρείται ότι το εμπόριο είναι εκτός του συστήματος που ισχύει σήμερα παγκόσμια, ενώ αντίθετα και το εμπόριο και η οικονομία και οι χρηματαγορές είναι άρρηκτα συνδεδεμένα σε εκφάνσεις της ε, παγκόσμιας οικονομίας. Ε, εξού και το γεγονός ότι οι σχετικές με τους τομείς αυτούς κρίσεις είναι αλληλένδετες. Γι' αυτό διαρθρωτικά θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ευθύνη των εμπορικών πολιτικών, των πολιτικών απελευθέρωσης όπως λέμε, φιλευθεροποίησης. Η διατροφική ας πούμε κρίση είναι κρίση που αφορά την αγορά α, τροφίμων, ε, η απερίμωση της υπαίθρου ε, είναι μια κρίση που αφορά την ε, πολιτική αστιφιλίας. Για το Καλιφόρουμ, ας πούμε, το είδαμε για την ΕΠΑ Καλιφόρουμ δεν συζητήσαμε το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Μιλήσαμε για την Κίνα, μιλήσαμε για την απελευθέρωση φιλοθροποίηση του τραπεζικού τομέα και ξέρουμε πόσο σημαντική σημαντικός είναι ο τομέας ε, στα πλαίσια τη κρίση. Το θέμα λοιπόν είναι πώ θα κάνουμε μια διάγνωση που δεν θα απομονώνει τις εκφάνσεις της κρίσης και κάθε τομέας θα λέει δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος τομέας. Και πώς θα διδαχθούμε τα διδάγματα αυτής της κρίσης ούτω ώστε η οικονομική κρίση ας πούμε των χρηματαγορών να μην οδηγήσει στο μέλλον σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Τέλος, λέτε στο εγγραφό σας ότι η Ντόχα μπορεί να είναι το σπιρούνι που θα δέσει νέα όθηση στην ανάκαμψη, στην αναπτυξία. Ήμουν στην ε, Ντόχα παλιότερα και άκουγα που λέγαμε ότι μετά το Σεπτέμβριο θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε συμφωνία ούτως ώστε να πάρει τα πάνω, του ή τα πάνω της παγκόσμια οικονομία. Αν είμαστε πεπισμένοι, όπως πιστεύω ότι είναι σωστό, ότι πρόκειται για μια διαρθρωτική κρίση, το θέμα δεν είναι ε, να αναζωπυρώσουμε την εμπιστοσύνη, ε, αλλά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στη ρίζα τους. Ω εκ τούτου το ερώτημα που απευθύνω στην Κομισιόν. Τι κάνουμε για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο ε, της οικονομικής ε, απελευθέρωσης και δύο, ποιο είναι το δίδαγμα που διδασκόμαστε και ενδεχομένω τρία ως ερώτημα προς τον Πρόεδρο αν μου επιτρέπει πώς δεδομένου του διαρθρωτικού και θα έλεγα συστημικού χαρακτήρα της κρίσης μπορούμε να ε, αξιολογήσουμε την κρίση ως τέτοια στο σύνολό της. Όχι οικονομική κρίση, όχι χρηματοοικονομική κρίση, όχι κοινωνική κρίση, όχι περιβαλλοντική κρίση μεμονωμένα, αλλά στο σύνολο, μια εγκάρσια δηλαδή θεώρηση των πραγμάτων. Ευχαριστώ. συμφωνώ απολύτως ότι χρειαζόμαστε μια συστημική προσέγγιση. Δεν πιστεύω όμως ότι απέχουμε πολύ από αυτή την προσέγγιση. Στο θεματολόγιο της ομάδας των G20 δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των διαφορών κρίσεων ή θεμάτων ή τομέων. Το περιβάλλον έχει ίση σε προτεραιότητα και σημασία θέση στο θεματολόγιο του G20 με την οικονομία ή την ενέργεια. Γιατί πάντα οι πολιτικοί άνδρες και οι γυναίκες, και αυτό βγήκε και από το Λονδίνο, είναι ότι όλες οι κρίσεις είναι τμήμα, όλες οι εκφάνσεις αν θέλετε της κρίσης, είναι τμήμα μιας συνολικής κατάστασης. Γι' αυτό πρέπει βεβαίως συνδεδεμένα να εξετάσουμε τα προβλήματα αυτά. Του συστήματος. Και υπάρχουν και καλά στοιχεία στο σύστημα, έτσι δεν υπάρχουν μόνο κακά. Το εμπόριο ας πούμε είναι από τα καλά στοιχεία του συστήματος, διότι υπάρχει ένα πολύ καλό σύστημα επίλυσης των διαφορών. Υπάρχει άμβλυνση, για να μην πω εξάλληψη των διαφορών μεταξύ των μικρών και μεγάλων ε, χωρών. Είναι αποτελεσματικοί οι κανόνες που ισχύουν. Σε μεγάλο βαθμό αποτρέπουν την ε, αναφύηση εκ νέου προστατευτισμού και σχετικών μέτρων Αλλά αν μια χώρα στα πλαίσια του ΠΟΕ αποφασίσει να πάει τους δασμούς της στο ανώτατο επίπεδο που επιτρέπει ο ΠΟΕ, θα έχουμε δισεκατομμύρια ε, σε απώλειες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν αρκεί η εφαρμογή των συμπεφωνημένων, αλλά πρέπει να έχουμε μια συνολική θεώρηση των πραγμάτων για να δούμε πώς σφαιρικά μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Και εμείς έχουμε μια πολύ ε, ολιστική προσέγγιση και περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες και ε, εξετάζουμε από την, ε, στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών θέματα βιωσιμότητας και είμαι πεπισμένος ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα Οπότε, επ' αυτή τη αγούση, οποιασδήποτε προτάσεις είναι καλοδεχούμενε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους λοιπούς ε, ομιλητές για τον προστατευτισμό. Συμφωνώ πλήρως με τον Ντέιβιντ. Τώρα υπάρχουν φαινόμενα όπως ε, ο έξυπνος, ο ευφυής προστατευτισμός ή ο και καλυμμένος. Να καταστήσω σαφές το εξής. Τον Ιούλιο, αν δεν απατώμε, η ετήσια έκθεση του ΠΟΕ, του 2009 δηλαδή, στην παρουσίαση αυτής της εκθέσεως, ο Πασκάλ Λαμή μας είπε ότι υπάρχει αναφύση νέων φαινομένων προστατευτισμού. Τώρα εσείς μας λέτε ότι τα πράγματα πηγαίνουν ε, καλύτερα. Άλλα λέει δε ο κλάδος. Το ερώτημά μου είναι μπορούμε να είμαστε ίσχυοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο θα προωθήσει το θέμα αυτό ή να ανησυχούμε ότι θα μείνουν τα πράγματα έτσι όπως είναι. Τώρα. Είπατε ότι η είσοδος στην κρίση ήταν συγχρονισμένη και αυτό σας έκανε εντύπωση. Ορθόν. Η έξοδος από την κρίση δεν θα είναι όμως συγχρονισμένη. Οπότε τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε, εφόσον θα υπάρξουν χώρες που θα βγουν από την κρίση νωρίτερα από άλλες. δεν θα πρέπει να σπρώξουμε τον ευρωπαϊκό κλάδο προς τις περιοχές εκείνες του κόσμου που θα εξέλθουν ταχύτερα της κρίσεως. Τέλος, για την ανάκαμψη. Είχαμε το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης. Έχουμε το Small Business Act προτίθεται η Κομισιόν να κάνει μελέτη αντικτύπου της εφαρμογής των μέτρων αυτών, διότι πέρασε ένας χρόνος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για την πρόσβαση στα κεφάλαια. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και θα πρέπει να τύχουν αξιολόγησης και εκτίμησης, διότι αφορούν άμεσα το εμπορικό δυναμικό της Ένωσης. Γιατί όταν μιλάμε για επιτυχή έξοδο από την κρίση, μιλάμε για επιτυχή έξοδο από την κρίση όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Και αν ξεχάσω κάποια απάντηση, θα προσπαθήσω να επανέλθω. Για τον προστατευτισμό. Το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία εξετάζουμε το θέμα ή τι απόχρωση προσδίδουμε στο θέμα. Αν κοιτάξουμε συγκεκριμένες χώρες, συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένες εταιρείε. Αν σταματήσουν οι εξαγωγές, ας πούμε, σε μια χώρα, ε, μπορεί να πλήξει τρομερά αυτό το μέτρο μία μικρομεσαία επιχείρηση παραδείγματος χάρη που εξαρτάται από εξαγωγές. Πρέπει να μειώσουμε τέτοιες ε, στάσεις. Γι' αυτό η Κομισιόν ε, πολύ γρήγορα ε, δημιούργησε ένα μηχανισμό παρατήρησης σε διμερές επίπεδο ε, και ένα μηχανισμό διαβουλεύσεων και κάθε φραγμός που θεωρείται διακριτικός, διακριτική μεταχείριση εντοπίζεται. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, παρακολουθούμε τα πράγματα τακτικά και λογοδοτούμε και στην Επιτροπή και στον ΠΟΕ. Νομίζω ότι όλα συνδέονται με ένα συστημικό τρόπο. Αυτό μοιάζει με τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα για το αντι Είναι σημαντικό το αντι αλλά αν δείτε το ποσοστό του εμπορίου που επηρεάζεται από το αντι-dumping είναι αμεληταίο. Το ίδιο μπορεί να υποθεί και για τις συνολικές παγκόσμιες εμπορικές ροές ε, και το πώς πλήττονται από τα μεμονωμένα προστατευτικά μέτρα. Δεν είναι σημαντική επίπτωση του προστατευτισμού στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Ακούμε δηλαδή από τη μία πολλούς να μιλούν για το προστατευτισμό ως σημαντική απειλή. Δεν είναι σημαντική απειλή, δεν είναι κίνδυνος, αλλά δεν πρέπει να επαναπαθούμε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πάνοπλοι. Επίσης, πέρα από τα γενικά θέματα, έχουμε και ειδικά θέματα που μπορεί να είναι πολύ σημαντικά και τα εξετάζουμε με κάθε σοβαρότητα. Ε, στο μήνυμα που δόθηκε από το G20 στο Pittsburgh, αυτό το σημείο ήταν πολύ σημαντικό και δεν θέλω να προδικάσω μια οποιαδήποτε επίσημη θέση που θα εκφράσει αυτές τις μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επαναλάβουμε την δέσμευση που ανελήφθη ε, στο ανακοινοθέν του G20 να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας να αναγνωρίσουμε τη σημασία του δηλαδή και να εντοπίσουμε το γεγονός ότι μόλις βγαίνουμε από την ύφαση, ύφεση αλλά δεν ξέρουμε πόσο στεναρή είναι αυτή η ανάκαμψη. Ε, θα πρέπει επίσης να σπρώξουμε το εμπόριο, τόσο ώστε να γίνει ατμομηχανή για την χρηματοοικονομική ανάκαμψη για το πώς θα βγούμε από την κρίση όλοι μαζί ή ο καθένας χώρια. Συζητείτε αυτό το θέμα και βλέπουμε στοιχεία α, ξεχωριστής χρονικής στιγμής α, εξόδου από την κρίση. Η ο καθενας χωρια συζητειτε αυτο το θεμα και βλεπουμε στοιχεια α ξεχωριστης χρονικης στιγμης εξοδου απο την κριση η κινα και οι αναδυόμενες οικονομίες ήδη έχουν περάσει σε θετικά νούμερα ανάπτυξης, ενώ εμείς ε, και οι αναπτυγμένε οικονομίε είμαστε σε αρνητικά επίπεδα ανάπτυξη. Και αυτό δείχνει ακριβώ ότι δεν βγαίνουμε όλη την ίδια χρονική στιγμή από την κρίση. Το να βγει επίσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν θετικά ε, στοιχεία, ας πούμε, ανάκαμψης για την ε, Γερμανία και τη Γαλλία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, Γερμανία και τη Γαλλία ως ατμομηχανή για να βγούμε και οι υπόλοιποι. Αλλά δεν, έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Η ανάκαμψη είναι άνηση και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και αυτό παραπέμπει πίσω στα δύο μηνύματα που ήθελα να σας πω. Τη σημασία της ενίας αγοράς και τη σημασία της διατήρησης των αγορών ανοιχτές. Είναι σημαντικό η, ευρωπαϊκή βιομηχανία να επωφεληθεί από την ανάκαμψη στην Κίνα και στην Ασία. Ε, και είναι σημαντικό η, ο ευρωπαϊκός κλάδος να έχει πρόσβαση σε φθηνές πρωτεσίλες για να υπάρχουν ανταγωνιστικές ε, εξαγωγές και αυτό να έχει ε, θετική επίπτωση με τη σειρά του στην ανάπτυξη. Επίσης, ε, η Κομισιόν έχει και το Small Business Act και άλλα συνοδευτικά μέτρα και στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ε, παρακολουθούμε τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης του εμπορίου, δεσμεύσεις που αναλύθησαν στο Λονδίνο. Πρέπει να δούμε όχι μόνο τις δεσμεύσεις βέβαια, αλλά και τη χρήση α, των ποσών αυτών, της χρηματοδότησης αυτής. Σε ποιο βαθμό δηλαδή, σε ποιο ποσοστό ε, γίνεται αίτηση ε, για χρησιμοποίηση κονδυλίων από διάφορες εταιρείε ε, για τη χρηματοδότηση εξαγωγών. Προσπαθούμε σε όλους αυτούς τους τομείς και σε άλλους τομείς να παίξουμε ενεργό ρόλο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το εμπόριο είναι θέμα της λύσης και όχι του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θαυμάσια παρουσίασή σας. Ε, και εγώ ίδιος έμεινα άναυδος. Ε, μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία για να προβληματιστούμε. Ε, μάλιστα σε μια συνεδρίαση που είχαμε οι συντονιστές ε, σκεφτόμαστε τι ακροάσεις ε, θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε και είχαμε σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κοινή ακρόαση με την ε, οίκων, με την ε, Επιτροπή δηλαδή Οικονομικών Υποθέσεων και με την Επιτροπή Εμπορίου, δηλαδή εμείς και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ε, να κάνουμε μια μεικτή ακρόαση, μια κοινή ακρόαση, νομίζω θα ήταν υποφελής για όλους μας. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στις αρχές του 2010. Σας ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε παρόντες.